Καλημέρα σας. Επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Λοιπόν, η πειθαρχία κάνει θαύματα αρκεί να την τηρούν όλοι. Σήμερα δυστυχώ δεν έχουμε φιλανδικά, θα ήθελα να σα ειδοποιήσω. πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ, ειδικά για όσου θέλετε να ακούσετε τώρα φιλανδικά. Αρχίζουμε.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 Κύριε εισηγητά, 12 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος ε, κατά. Η κυρία Πιτέρα δεν έχει μαζί την κάρτα τη δεν πειράζει όμω. Ωραία. Τελείωσε αυτό το θέμα. Επόμενο, 8. Τώρα καλό θα ήταν να είχαμε και κανέναν επίτροπο παρόντα. Πού είναι ο κύριος επίτροπος? Genau, kann mal jemand vor der Tür betreiben. Μπορεί να στείλουμε, να στείλουμε κανένα ανοιχνευτή τώρα έξω από την αίθουσα, βρούμε πού είναι ο Επίτροπος. Genau. Genau. Jedenfalls möchte ich Sie herzlich das zuständige Θέλω να καλωσορίσω θερμά, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Μιλιώνη, αρμόδιο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Θα καταφτάσει ο, ο Επίτροπος, όπως και ο εισηγητή, φαντάζομαι. Αλλά ειλικρινά έχουμε εδώ κόσμο που περιμένει. Και ο χρόνος αναμονής είναι χρόνος από τη ζωή μας. Λοιπόν, θα αρχίσουμε μόλις έρθει ο κύριο Χόγκαν.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 Stress soll ja auch gesund sein, von daher. Tut mir leid, also. Ja, it's, it's as, as every day, but we know it beforehand. Καλά κίνηση έχει κάθε μέρα, τι να κάνουμε, τα ξέρουμε αυτά. Yeah. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, αλλά πραγματικά έχω μπουχτήσει Πάντα περιμένουμε κάποιον άλλη συνεδρίαση. Και χαιρόμαστε που είχε έρθει το ελεκτικό συνέδριο, που έρχεται από τόσο μακριά. Πιο μακριά από όλους είναι το ελεκτικό συνέδριο, αλλά είναι εδώ. Ζήτω, ήρθε και ο Επίτροπος, καλώς ορίσατε. it's a, it's a, it's a kind of strategy to put you a little bit under stress. Και αυτό στρατηγική είναι να μας τρεσάρετε λίγο, να μας πρεσάρετε. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 8. Συνεχίζουμε το σημείο 8, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καλωσορίζω θερμά τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Χόγαν. Καλωσορίζω και τον Γενικό Διευθυντή και γενικότερα τη Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε επίτροπε. Ε, ε, κύριε Πλεύρα, είναι εξαιρετική έκθεση πεπραγμένων ε, με ιδιαίτερη χαρά. Ευχαρίστηση τα διαβάζει κανείς και γνωρίζουμε, ε, ξέρουμε να τα εκτιμάμε αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιό μας και για την προθυμία να έρθετε να ανταλλάξουμε απόψεις. Κύριε Πίτροπε, μόλις ξέρετε τι έχετε να πείτε, μπορείτε να πάρετε μέσα στο λόγο. Α, όχι, ο κύριος Μιλιώνης. Κύριε Μιλιώνη, παρακαλώ, εσείς πρώτα. Παρακαλώ. Τώρα το περιμέναμε τόση ώρα γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα των εργασιών ε, δήλωσης ε, διασφάλισης του ελεκτικού συνεδρίου για τους φυσικούς πόρους σήμερα. Ε, το 2016 εκτιμήσαμε το επίπεδο ασφάλματος στο 2,5% για τον τομέα φυσική πόρη στο σύνολό τους. Το νούμερο αυτό είναι πάνω από το κατόφλιο σημαντικότητα στο 2% αλλά κάτω από την εκτίμηση του περσινού έτους του 2,9%. Επιπλέον έχουμε δύο επιμέρους αξιολογήσεις, μία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Γεωργικών Εγγυήσεων ε, υποστήριξη αγορά και άμεσες ενισχύσει και ένα για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κλιματική δράση και την αλία. Και το μεγαλύτερο επίπεδο σφάλματος ήταν στο δεύτερο τομέα. Το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κλιματική δράση και την αλία παραμένει στο 4,9% πάνω από τη σημαντικότητα, αλλά ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμησή μας για πέρυσι 5,3%. Σε 16 περιπτώσεις βρήκαμε ότι οι εθνικές αρχές είχαν επαρκείς πληροφορίες για να ανεχνεύσουν τα σφάλματα. Αν αποφεύγαμε το επίπεδο σφαλμάτων ε, θα, είχε, θα ήταν διαφορετικό κατά, 1,5, ε, κατά μία μισή ποσοστία μονάδα. Όπως τα περασμένα ε, χρόνια τα έργα που σχετίζονται με επενδυτικά θέματα αφορούσαν το 60% του εκτιμόμενου επεδοσφάλματος σε σύγκριση με το 1 τρίτο των σφαλμάτων που σχετίζονται με το ΜΙΣ. Φέτος, τρία από τα μεγαλύτερα σφάλματα επιλεξιμότητας περιλάμβαναν δικαιούχους που είτε δεν αποκάλυψαν ότι ελέγχονταν είτε ε, είχαν επαφέ με συνδεδεμένε εταιρείε, παραβιάζοντα του ε, ευρωπαϊκού και εθνικού κανόνε. Συνιστούμε λοιπόν η Κομισιό να δώσει οδηγίε ε, για βέλτιστε πρακτικέ μέσω νέων τεχνολογιών πληροφορική, για παράδειγμα, μεταξύ εθνικών αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι θα εντοπίσουν συνδέσει μεταξύ ετούντων και λοιπόν ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στα αναφερόμενα έργα. Τώρα, όσον αφορά τις άλλε δευτερεύουσες αξιολογήσει του EAGF αγορά και άμεση ενίσχυση, το εκτιμόμενο επίπεδο σφαλματός μα είναι στο 1,7%. Το ποσοστό αυτό είναι κάτω από το κατόφλιο σημαντικότητα του 2% και αντιστοιχεί σε βελτίωση σε σύγκριση με την περσινή τιμή του 2,2%. Το EAGF αντιστοιχεί σε πάνω από τα 3 τέταρτα των σχεδόν 58 δισεκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν στο πλαίσιο του τομέα 2 φυσική πόρη του MFF. Ε, ε, Ξέρουμε ότι υπάρχουν λιγότερα ασφάλματα λόγω υπερβολικής δήλωσης, υπερβολικά δηλωμένης ή ε, μη επιλέξιμης γης για τις οποίες έχουν θέσει αξιώσεις οι γεωργοί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βρει τεράστια ασφάλματα όσον αφορά τον καθορισμό του μόνιμου λιμώνα. Τώρα φαίνεται να έχει διορθωθεί η κατάσταση χάρη σε, μια, σε ένα νέο πιο ευέλικτο καθορισμό του μόνιμου λιμώνα. Τα σχέδια δράσης ε, έχουν επίσης βελτιώσει τα δεδομένα στα LPIS και με το νέο γεωχωρικό σύστημα online ε, υποβολής των αιτήσεων και αυτό έχει βοηθήσει στη βελτίωση. Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που ελέγξαμε τη συμμόρφωση των νέων υποχρεώσεων greening για τους ε, γεωργούς ε, που είχαν οδηγήσει σε πολλά ασφάλματα. Ε, τα ασφάλματα που διαπιστώσαμε σχετίζονταν κυρίως με τις απαιτήσει για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, τις EFA. Επίσης βρήκαμε αδυναμίες στην προστασία των μόνιμων λιμώνων. Η αρρώσιμη γη θα πρέπει να γίνει μόνιμη, μόνιμος λιμώνας εφόσον θα θεωρείται μόνιμος λιμόνας εφόσον έχει καλυφθεί με χορτάρι για πέντε ε, συνεχή χρόνια. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν είχαν ιστορικά δεδομένα ελέγχου της μόρφωσης ε, αυτόματα με αυτή την υποχρέωση. Αλλά κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ταξινομήσει αξιόπιστα το μόνιμο λιμόνα. Συνιστούμε λοιπόν η Κομισιόν να αναθεωρήσει την προσέγγιση των χρηματοδοτικών οργανισμών όσον αφορά την κατηγοριοποίηση και την επικαιροποίηση των κατηγοριών γης ε, στο ε, LPIS και να πραγματοποιήσουν διασταυρούμενους ελέγχους. Επίσης βρήκαμε ότι 63 αγροκτήματα που επισκεφθήκαμε συμμορφώνονταν με την διαφοροποίηση καλλιεργιών. Όσον αφορά τα μέτρα αγοράς, παρότι ε, αντιστοιχούν σε μικρό κομμάτι του συνολικής δαπάνης EGF, τα σφάλματα που βρήκαμε αποτελούν σημαντική ε, πηγή υπερβολικών ε, πληρωμών για το Ταμείο στο δείγμα μας. Στην έκθεση ετήσιων δραστηριοτήτων της, η DJ Agri παρουσιάζει συνολικό προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος ε, για τις δαπάνες της ΚΑΠ στο 2,5%. Κάτι που συνάδει με τη δική μας εκτίμηση. Το ποσοστό αυτό βασίζεται σε συνολικό επίπεδο σφάλματος 1,2% όπως αναφέρουν τα κράτη-μέλη, στο οποίο προσαρμόζει η Κομισιόν βάση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και σε μικρότερο βαθμό ε, στις γνωμοδοτήσει των οργανισμών πιστοποίησης. Σε μια ειδική έκθεση για τα σώματα ε, για του οργανισμού πιστοποίηση που δημοσιεύτηκαν φέτο, κάναμε διάφορε συστάσει για βελτιώσει που θα συμπεριληφθούν στι νέε κατευθυντήριε γραμμέ τη Κομισιόν από το οικονομικό του 2018 και μετά. Επίσης έχουμε καλύψει ζητήματα επιδόσεων της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής. Αυτό το πρώτο έτος του greening χρησιμοποίησαμε το δείγμα για την ε, ε, δήλωση αξιοπιστίας ε, για τις νέες ε, πρακτικές γεωργίας. Επισκεφτήκαμε 197 αγροκτήματα, όπου διαπιστώσαμε ότι το 11% χρειάστηκε να αυξήσει την διαφοροποίηση καλλιεργιών και το 32% έπρεπε να αυξήσει τους ε, χώρους οικολογικής εστίασης, τις περιοχές οικολογικής εστίασης. Αυτό επηρέασε το 3,5% περίπου της αρρώσιμης γης των, ε, του δείγματο αγροκτημάτων. Ε, σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε σε δύο εβδομάδε μια ειδική έκθεση για το σχεδιασμό και το πρώτο έτο υλοποίηση του Greening το 2018. Την τελευταία τριετία έχουμε πραγμα... εξετάσει ζητήματα επιδόσεων για ένα δείγμα συναλλαγών αγροτικής ανάπτυξης. Το 95% των έργων που συμπληρώθηκαν που ολοκληρώθηκαν την εποχή του ελέγχου μας ε, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο. Αλλά περίπου στο 1 τρίτο των περιπτώσεων, 34% δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ότι τα κόστη ήταν εύλογα. Η χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστου έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τον κίνδυνο υπερβολικών τιμών. Σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε μια έκθεση για αυτό το ζήτημα το 2018. Επιπλέον, για να κλείσω, θα μιλήσω για τους τομείς όπου χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Ε, η πρόοδος χρειάζεται χρόνο για να επιτευχθεί όπως αποδεικνύεται. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Με νέες ειδήσει και παλαιότερες. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που μου προσφέρετε να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε την γεωργική πολιτική. Τα αποτέλεσματα δείχνουν φέτος ότι η ΚΑΠ εξακολουθεί να προσθέτει αξία διασφαλίζοντας ε, υγιείς και κανονικές δαπάνες. Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση είμαι ικανοποιημένος το Ελεκτικό συνέδριο και οι Κομισιόν έχουν συμφωνήσει για το ποσοστό σφάλματος 2,5% κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Ε, αυτό είναι από τα θετικά μηνύματα από τα συμπεράσματα του Ελεκτικού συναδρίου, ότι δεν υπάρχουν υλικά ασφάλματα, ότι στην αγροτική ανάπτυξη το ποσοστό ασφάλματος εξακολουθεί να μειώνεται και έχει δώσει ε, για πρώτη φορά θετική γνωμοδότηση το ελεκτικό συνέδριο από το 1994. Μπορούμε να βλέπουμε πολύ θετικά και μεγάλη περηφάνεια τα αποτέλεσματα αυτά. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι το 2016 ήταν το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής της ε, μεταρρύθμισης ε, και των πυλώνων 1 και 2. Οι άμεσες ενισχύσεις για πρώτη φορά ακολούθησαν τους νέους κανόνες και στην Κομισιόν εξακολουθούμε να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες φάλματος και να προτείνουμε συστημικές λύσεις. Τα κράτη-μέλη επένδυσαν χρήμα και χρόνο για την επικαιροποίηση και τη διαχείριση των νέων συστημάτων ελέγχου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μη επιλέξιμοι μόνιμοι λιμόνες ε, υπήρχαν, ήταν ανέκαθεν πηγές ασφαλμάτων. Ε, Σήμερα πλέον αυτό δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Με τον αναθεωρισμένο ορισμό του μόνιμου λιμώνα που εισήχθη με την μετρήθμιση του 2013 ε, διευκολύνθηκε η επιλεξιμότητα. Ταυτόχρονα βελτιώθηκε και η εξοπιστία των δεδομένων στα συστήματα. Φυσικά αυτό συμβαίνει για τι ε, ενισχύσει που βασίζονται σε περιοχέ. Η κατάσταση για την αγροτική ανάπτυξη είναι πιο περίπλοκη. Έχουμε επιτύχει πολλά σε θέματα επιδόσεων εκεί και ενώ πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε. πρέπει επίση να αφήσουμε χρόνο ώστε κάποιε πρωτοβουλίε μα να φέρουν αποτελέσματα και να τηρήσουμε τους στόχους μας αντί να φτιάχνουμε νέες πρωτοβουλίες. Τα συνολικά συμπεράσματα είναι ότι το ποσοστό ασφάλματος είναι χαμηλό και τα χρήματα έχουν δαπανηθεί με υγιή τρόπο για τι μεταρρυθμίσει, Οι μεταρρυθμίσει τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά. Οι νέε ενισχύσει λειτουργούν. Καλύπτει το 77% τη ε, γεωργική γης. Είναι η πρώτη φορά που ένα σύστημα ε, υλοποιείται με τόσο ευρία κάλυψη, όχι μόνο για την παραγωγή, αλλά για περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Είναι ήδη σαφέ ε, ότι οι αγροτικές πρακτικές επηρεάζονται από τι νέε απαιτήσει. Το 14% τη αρρώσιμη γη έχει δηλωθεί ω γη οικολογική εστίαση πολύ ψηλά πάνω από το υποχρεωτικό 5% κάτι που αυξάνει τη θετικά αποτελέσματα για τη βιοπικιλότητα. Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν σχεδόν άψογη, άψογο ποσοστό απορρόφησης 97% ε, απορροφήθηκε το 2016 με ακόμα ε, υψηλότερο ποσοστό 98% το 2017 η αγροτική ανάπτυξη. Πάνω από το 20% έχει ήδη δαπανηθεί ε, ποσό 21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα περισσότερα παλιά προγράμματα έχουν κλείσει με απορρόφηση 99% των διαθέσιμων κονδυλίων. Τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με τα παλιά προγράμματα δηλαδή από το 2007 μέχρι το 2013, θα αποτελέσει το αντικείμενο εκθέση μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Τι γίνεται ε, με την ΚΑΠ τώρα ε, σε φάση υλοποίηση. Το 2015 και 2016 ήταν δύσκολα χρόνια, ειδικότερα ε, για τα γαλακτοκομικά και το χείριο κρέα. Η Κομισιόν υποστήριξε του τομεί αυτού αναγνωρίζοντα τι δυσκολίε. Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ διατέθηκαν προ υποστήριξη του και των δύο τομέων το 2015. Ω αποτέλεσμα των δράσεων τη Κομισιόν και τη υποστήριξη προ τον τομέα έχουμε σαφή ενδείξει ανάκαμψη το 2016. Η αγορά κρέατο έχει ανακάμψει ε, σαφώς πέρυσι με καλύτερες τιμές για τους γεωργού ε, και καλύτερη ισορροπία προσφορά και ζήτηση. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο ε, ένα βιώσιμο μέλλον για τον τομέα και για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτόν ώστε η αντοχή τους και η αντοχή των μεθόδων παραγωγή να βελτιωθούν. Αυτό θα το εξετάσουμε βάσει της ανακοίνωσης της Κομισιόν για το μέλλον ε, των τροφίμων και της ε, γεωργίας που θα ε, εμφανιστεί αύριο. Βιώσιμο μέλλον σημαίνει νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, προσέλξη νέων ανθρώπων και καινοτομία. Η γεωργία αποτελεί κλειδί για τις γεωργικές μας περιοχές. Είναι ένα τομέα που αξίζει κάποια προστασία από τις πίεσεις της αγοράς. Υποστηρίζω λοιπόν τις άμεσες ενισχύσεις για να διασφαλιστεί βασικό εισόδημα για τους γεωργούς μας και σταθερότητα όσον αφορά την απασχόληση. Συμφωνώ ωστόσο ότι πρέπει να είναι δίκαιες και να αφορούν πραγματικούς γεωργούς. Γι' αυτό το λόγο η μεταρρύθμιση του 2013 περιλαμβάνει πολλές διατάξεις ε, ε, για τη σωστή κατανομή των πληρωμών, αυτό περιλαμβάνει διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων το εθελοντικό ανώτατο όριο. Μπορούν να γίνουν περισσότερα, αλλά αυτό θα γίνουν μετά το 2020 και θα συζητήσουμε διάφορες λύσεις πολύ σύντομα, είμαι βέβαιος. Στην τωρινή προγραμματική περίοδο Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 125.000 νέε θέσει εργασία, 60.000 νέε αναδυόμενε νοφεί επιχειρήσει. Έχει γίνει ήδη σημαντική πρόοδο. Οι επενδύσει αυτέ θα διαφοροποιήσουν την αγορά θέσεων εργασία και θα βελτιώσουν την πρόσβαση στι υπηρεσίε που είναι περιορισμένε στι αγροτικέ περιοχέ. Έτσι θα προσελκυθούν ε, περισσότεροι νέοι άνθρωποι ε, στη γεωργία και θα διασφαλιστεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, το βιώσιμο μέλλον σημαίνει επίσης ε, προφύλαξη των φυσικών πόρων. Ήδη τα νούμερα είναι ενθαρρυντικά. 24% μείωση των ε, επιβλαβών ε, εκπομπών, 18% μείωση των νητρικού άλατος στα ποτάμια και σημαντικές βελτιώσεις γενικά κλιματικές τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ ε, θα περιλαμβάνουν μια σοβαρή δέσμευση για περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Αυτό ικανοποιεί και τις προσδοκίες ε, των λαών μας ε, όπως ε, διαφαίνεται στην ε, δημόσια διαβούλευση που κάναμε νωρίτερα φέτο. Στο διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν είναι μόνο πράσινη και βιώσιμη αλλά και ανταγωνιστική και δίκαιη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέα ε, της Γεωργίας ε, παγκοσμίω προσφέρει σωστέ τιμέ. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση των εξαγωγών. 130 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι η κύριοι εισαγωγή ε, είναι η ΙΠΑ, η Κίνα και η Ελβετία. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ε, αγροδιατροφικών προϊόντων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, εισαγωγές που ανέρχονται στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 και το 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι ένας υπεύθυνος εμπορικός εταίρος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διασφαλίζουμε με τους εταίρους μας στην Αφρική ότι θα υπάρξουν υπεύθυνε επενδύσεις ε, στην Αφρικανική Γεωργία. Τα περισσότερα προστατευτικά μέτρα της ΚΑΠΑ ε, βοηθούν στη σταθεροποίηση της αγοράς ε, και ευνοούν τις εισαγωγές. Οπότε βρισκόμαστε ε, στην πρώτη γραμμή ανάπτυξη της γεωργίας στην Αφρική. Υποστηρίζουμε την έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη προτύπων, τη βιολογική παραγωγή και ταυτόχρονα πολλές από τις φτωχές χώρες έχουν σοβαρέ ελλείψει σε γαλακτοκομικά, με προϊόντα όπω το γάλα, τα οποία μπορούν να καλυφθούν μόνο από τι εισαγωγέ. Οπότε με τα νέα μα ΚΑΠ δεν χρειάζονται πλέον να φοβούνται για ελλείψει. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη έχει βιώσει βιώσιμη γεωργία, διασφαλίζει ε, τις ε, τροφίμων στην ποιότητα που επιθυμεί ο κόσμος ε, αυτό με ισορροπία όσον αφορά τα εισοδήματα των γεωργών μας. Θέλουμε να σχεδιάσουμε έξυπνα και αποτελεσματικά για το μέλλον την πολιτική αυτή. Υπάρχουν ήδη πρακτικές σε κράτη-μέλη και να δαπανώνουμε τους τον προπολογισμό μας με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο. Χαίρομαι που διαπιστώνεται και επικυρώνεται από το ελεκτικό συνεδρίο ότι η διαχείριση γίνεται, η διαχείριση γίνεται σωστά, ότι τα αποτελέσματα αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικά και ότι τα κράτη-μέλη έχουν καταφέρει ε, τόσο πολλά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε νέα βήματα στο μέλλον, να εστιαστούμε στι επιδόσει. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι και να σα διαβεβαιώσω και πάλι ότι ο οποιοδήποτε σχεδιασμό μελλοντική πολιτική θα πρέπει να βασιστεί στι στιβαρέ δομέ που ήδη υπάρχουν για την ΚΑΠ, ώστε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε θα ήθελα να πω το εξή για την Επίτροπή μας. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, η αγροτική ανάπτυξη, είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρεται ρητά. Στις έκτακτες ε, εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, βλέπουμε ότι όσο πιο δυσμενής είναι, τόσο πιο χαμηλό βαθμός είναι ο υπάλληλος που το χειρίζεται αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μη στέλνετε ε, τμήματάρχε ή αναπληρωτέ, Δεν είναι δίκαιο κάτι τέτοιο. Στην τελευταία έκθεση το 2017 για την αγροτική ανάπτυξη διακόψαμε τις συζητήσει γιατί είναι άδικο. Και σήμερα θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σα. Το λόγο τώρα έχει εισηγηθεί ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο για την ετήσια έκθεσή του για τη χορήγηση απαλλαγή στον προπολογισμό. Όπως πάντα, για μας αυτή είναι η βασικότερη ε, έκθεση για την εργασία μας, για να εκπονήσουμε την έκθεση τη δική μας για την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χόγκαν και τους συνεργάτες του και για τη δική τους ετήσια έκθεση, αλλά και πιο πρόσφατα για τις εκτενείς απαντήσεις στις περισσότερες από 40 γραπτές ερωτήσεις που υποβάλαμε. Η Γεωργία πάντα κυριαρχεί στο επίκεντρο της προσοχής ε, του προϋπολογισμού ε, και της απαλλαγής, γιατί είναι το 40% των πόρων που ε, απόρροφα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει όλη μας την προσοχή γιατί είναι και ιδιαίτερη περίπτωση. Ωστόσο, η απαλλαγή δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μια υπόθεση αριθμών και στοιχείων και δεδομένων. Αλλά σκοπό έχει να αξιολογήσουμε κιόλα κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στους στόχους που είχαμε θέσει για την κοινή γεωργική πολιτική. Οι πολιτικές αξιολογήσεις είναι αυτές που πρέπει να γίνουν και να ρωτήσουμε έχει καμία προστιθέμενη αξία και ποια η κοινή γεωργική πολιτική σε σχέση και με τους διατηθέμενους πόρους. Αυτό ισχύει για τη μελλοντική εκπόνηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Την έχουμε μπροστά μας ακόμα αυτή τη συζήτηση και πρόκειται να γίνει. Όπου θα κυριαρχήσει και αυτό το θέμα και θα επηρεάσει τη μελλοντική κατανομή των πόρων. Όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξόδου ε, μιας από τις μεγαλύτερες ε, συνεισφέρουσες χώρες. Πράγμα που θα κάνει τη συζήτηση ακόμα πιο συναρπαστική. Ένα είναι γεγονός. Είναι πολλές επιφυλάξεις και ε, τα ρίσκα που συνδέονται με κάποιες δαπάνες, γιατί υπάρχουν οι κανόνες, όπως είναι το πρασίνισμα, το greening, το τόνισε και το ελεκτικό συνέδριο αυτό. Ε, εδώ το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει μεν ε, ήδη μεγάλη βελτίωση, αναμένεται ειδική έκθεση την οποία έχετε ανακοινώσει και την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει αύξηση του αριθμού σφαλμάτων στον πρώτο πυλώνα, αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο ε, της τάξεως ε, από το 1,38% μέχρι 1,96%. Τρεις θέσεις, τρία ψηφία μετά την υποδιαστολή ε, παραμένει κάτω του στατιστικού σφάλματος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Σταθεροποίηση 4% στην αγροτική ανάπτυξη των σφαλμάτων. Εδώ παραμένουμε πολύ ψηλότερα από το στατιστικό λάθος. Πώς θα βελτιωθεί αυτό. Υπάρχουν διάφορα μέτρα, αλλά είναι πολύ διαφορετικοί φορείς που τα χειρίζονται αυτά στα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να μειωθεί το ποσοστό αυτό σφάλματος. Και πάλι περιμένουμε ενδιαφέρον αλλά και το 4% ε, καλή τιμή είναι. Για τα μέτρα για την αγορά βλέπουμε 2,85% μείωση. Ε, το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει 1,7% σφάλμα για τον πρώτο πυλώνα και ελαφρά βελτίωση στην αγροτική ανάπτυξη 4,9%. Άρα στο πρώτο πυλώνα βρισκόμαστε κάτω από τις διαπιστώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Στην αγροτική ανάπτυξη δεν συμφωνεί πάρα πολύ, είναι λίγο παραπάνω, αλλά σαφής βελτίωση από το 2015. 2,5% του συνολικού σφάλμα, εδώ συμφωνούν Ελεκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι σαν να συνήθιστο ο ελεγκτή και ο ελεγχόμενο να καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τώρα, τι διδάγματα βγάζουμε εμείς από τους αριθμούς αυτούς, επανειλημμένα το έχουμε ακούσει, το λεγόμενο πρασίνισμα. Κύριε Επίτροπε, εσείς διαπιστώσατε ότι οι συνάδελφοι εδώ της Επίτροπη έκαναν πολλές ερωτήσεις σχετικά και στην ετήσια έκθεση του το ελεκτικό συνέδριο μας έκανε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το greening. Σας είπα, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την ειδική έκθεση για το greening. Αυτή τη φορά συμφωνούν Ελεκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα είναι περίπλοκο βέβαια του πρασινίσματος. Από τη μια έχουμε στάνταρ μέτρα για τη διαφοροποίηση ε, των ε, καλλιεργειών, για τους μόνιμους βοσκοτόπους και μόνιμους λιμόνες και μέτρα για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κράτη-μέλη και επιτόπου ε, φορείς και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι το θεωρούν υπερβολική επιβάρυνση. ισχύει ακόμα το παλιό σύστημα εντός εισαγωγικών της ε, πολλαπλής συμμόρφωσης και από εκεί και πέρα έχουμε τρία διαφορετικά συστήματα με διαφορετικά διοικητικά εργαλεία. Ε, εκφράστηκε μια επιθυμία για απλούστευση. Δεν ανταποκρίνονται όλα αυτά στην απλούστευση όμως. Και πιστεύω ότι και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής γεωρικής πολιτικής χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών. Θέλω να επιμείνω λίγο στην προστιθέμενη αξία της, ε, του προσυνήματος. Στο έγγραφο εργασίας στο υπηρεσιακό του 2016 ορίζεται και παραθέτω στα αγγλικά. Γενικά οι αγρότες θα πρέπει να αλλάξουν καλλιέργεια ε, λιγότερο από 1% για να έχουμε διαφοροποίηση και ε, και να ανταποκριθούμε. Και είναι πρακτική που ακολουθούν οι αγρότες οι οποίοι ήδη συμμορφώνονται ε, γιατί οι αγρότες καλλιέργειες καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια ε, και στη σελίδα 9 εξαρτάται αυτό σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές των κρατών μελών και των αγροτών. Ε, λίγα είναι τα κράτη-μέλη που φιλοδοξούν να περιορίσουν στους περιοχές οικολογικής συστίασης, στη χρήση ζανιοκτώνων και ε, φυτοφαρμάκων. Σε ό,τι αφορά αυτές τις περιοχές οικολογιστής εστίασης και πάλι περιμένουμε την έκθεση του ελεκτρικού συνεδρίου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα Ελεκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό ότι η διαφοροποίηση και τα νέα μέτρα δεν έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές ε, στις ε, εκτροφές και στις ε, επιχειρήσεις που επισκεφτήκατε. Στο πρώτο πυλώνα δεν έχουμε πρόβλημα συμμόρφωσης αλλά επιδόσεων ε, και θα πρέπει να προσανατολιστούμε περισσότερο στις επιδόσεις και λιγότερο στη συμμόρφωση. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το compliance αλλά το performance. Ε, Επίση υπάρχει και ένα πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ε, που δεν έχει ε, αποφέρει ακόμα τους επιθυμητούς καρπούς και το ε, πρασένισμα μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες στην κατανομή των πόρων μεταξύ των αγροτών εάν δεν υπάρχει η ε, δίκαιη μεταχείριση. Δύο λόγια για την αξιοπιστία των δεδομένων που δίνουν τα κράτη-μέλη. Κύριε Επίτροπε, είδατε στι γραπτέ ερωτήσει ότι ανησυχούν τα μέλη τη Επιτροπή μα για την ποιότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων των κρατών μελών. Η Γενική Διεύθυνση Άγκρη ε, έκανε 52 top-ups, 32 ε, προσαρμογές ε, και 39 στην αγροτική ανάπτυξη. Οι περισσότερες προσαρμογές όμως αφορούσαν ε, ποσά και ποστό κάτω του 1%. Άρα είναι περιορισμένο. Για τους δείκτες κλειδιά και την δίκαιη κατανομή και τον επιμερισμό των πόρων. Στην τελευταία μας έκθεση είχαμε αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο ε, το 80% των δικαιούχων να παίρνουν 20% των πληρωμών και το 44% των εκμεταλλεύσεων να εμφανίζουν τζίρο κάτω των 4.000 ευρώ ετησίως. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Κάτι τρέχει με την κατανομή των πόρων. Αρκεί να κοιτάξει κανείς αυτά τα στοιχεία για να καταλάβει ότι οι μεγάλοι οι οποίοι έτσι κι έχουν κερδοφορία παίρνουν περισσότερα. Ενώ οι πολύ μικροί αγρότε που είναι στα όρια της επιβίωσης δεν ε, ανήκουν στους δικαιούχους. Πόσο μάλλον στην έκθεση δραστηριοτήτων βλέπουμε ότι το 51% ε, των δικαιούχων των αμέσων πληρωμών παίρνουν κάτω των 1.250 ε, ευρώ έκαστος, δηλαδή κάτω από 4% του συνόλου. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά ας μας επιτραπεί το ερώτημα για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, προτείνει, για να μην πω επιβάλλει τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο και τι προτίθεται να κάνει στο μέλλον έτσι ώστε να διορθωθούν αυτά τα κακό κείμενα. Διότι ακούγονται και φωνές όλο και περισσότερο ότι στην κατανομή των γεωργικών πόρων θέλετε να προχωρήσετε διαφορετικά. Αν δω τι γίνεται στη Γερμανία και συνολικά στην Ανατολική Γερμανία αλλάζουν χέρια υγιές, αγοράζουν ε, πολλές yes, επενδυτικά ταμεία, επενδυτές, εταιρείες και γεωργικές γεές και δάση ε, και φαίνεται ότι η γεωργία και η δασοκομεία πλέον είναι επένδυση ε, για να τοποθετήσει κανείς τα χρήματά του και να έχει καλή απόδοση. Δεν έχει σχέση με τη γεωργία πλέον. και υπάρχει μια τάση ε, για εκβιομηχάνηση τη Γεωργία. Αυτά που δεν κατάφερε η ΤΕΤΕΡ, η Ανατολική Γερμανία και ο σοσιαλισμό, φαίνεται τα καταφέρνει τώρα ο καπιταλισμό και η νέα οικονομία. Και δεν ξέρω, αυτό είναι το οποίο που θέλουμε να δούμε στο μέλλον. Εγώ ταξιδεύω πολύ εκεί και διανύω χιλιόμετρα και βλέπω δεξιά και αριστερά καλλιέργειες ε, ε, ε, του για παραγωγή βιομάζας. Δηλαδή είναι βιομηχανική γεωργία. Στον κανονισμό Omnibus προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρεθεί έννοια του ενεργού αγρότη. Αυτό προτείνει και η Ένωση Γεωργών από το Βραδεβούργο. Δηλαδή να ενισχύονται αγρότες ντόπιοι που ασχολούνται με τη γεωργία κατά κύριο επάγγελμα και στο μέλλον κάποιες εταιρείες με ανώνυμους ή απρόσωπους ιδιοκτήτες, με επενδυτικές ε, εταιρείες, να μην θεωρούνται αγρότες και να παίρνουν και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια γεωργία θέλουμε πρέπει να αλλάξουμε τακτική και πραγματικά επιδοτήσει και βοήθειε να πηγαίνουν σε εκείνου που ε, χρειάζονται τα χρήματα, που εργάζονται, που καλλιεργούν τη γη του και δεν ε, κερδοσκοπούν. Και ε, φροντίζουν την παραδοσιακή και αηφόρο και βιώσιμη γεωργία. Στην ίδια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για τους νέους αγρότες να καταβάλλονται οι πληρωμές μετά από την, τον έλεγχο των όρων χρειάζεται κάποια ευελιξία στον ορισμό του μόνιμου λιμώνα ή βοσκοτόπου, αλλά θεωρεί σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν ε, ότι πρέπει να το επεκτείνει σε οτιδήποτε χρησιμοποιείται για βοσκή. Μπορεί να είναι ε, θαμνώδεις εκτάσεις μέχρι και δασικές. Ε, επόμενη ερώτηση. Η φετινή απαλλαγή, κύριε Επίτροπε. είναι η τελευταία ευκαιρία να δούμε τι θα κάνουμε πριν τι διαπραγματεύσει για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επειδή είμαι μέλο και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε εάν ισχύει αυτό που ακούμε για την αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς τρίτες χώρες είναι εις βάρος της ντόπια γεωργίας εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αφρική ακούμε ότι καταστρέφουμε τη γεωργία γιατί με επιδοτούμενα προϊόντα που εξάγουμε είμαστε πιο φτηνοί σε σχέση με τους ντόπιου παραγωγούς ε, και είναι εκτός ανταγωνισμού ξέρω ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενισχύσεις εξαγωγικές αλλά τα προϊόντα αυτά καθ' αυτά όταν επιδοτούνται ε, είναι φθηνότερα. Έχουμε πάντα ε, το επιχείρημα ότι επειδή χάθηκε η ρώσικη αγορά ε, επιβαρύνονται οι γεωργικές επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται τις ίους εξαγωγές. Και έχουν βρεθεί και άλλοι τρόποι να παρακάμπτεται αυτό με την Τελωνιακή Ένωση μέσω τρίτων κρατών. Εξ όσων γνωρίζω. Και φτάνουν μέχρι και στη Ρωσία ευρωπαϊκά προϊόντα πλαγίως. Δίκαιη κατανομή λοιπόν των πόρων ε, στάνταρ για το περιβάλλον, ενίσχυση των νέων αγροτών. Όλα αυτή είναι η κοινή δεδηλωμένη μα στόχη και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Ζέλερ. Να επαναλάβω αυτά που εσείς κυρία Πρόεδρε ε, και ο κύριος Ζέλερ αναφέρατε ότι πρέπει δηλαδή να παρακολουθούμε πολύ στενά το τι συμβαίνει στην έκθεση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και όταν το νούμερο μειώνεται, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε αυτό. Και βεβαίω θα λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσατε σε σχέση με τι προμήθειε και τα project που εξελίσσονται και όπου τα κράτη-μέλη μας υποδεικνύουν περίπλοκες καταστάσεις όπου οδηγούμαστε σε σφάλμα. Αυτά θα τα λάβουμε υπόψη στη διαδικασία των νομοθετικών αλλαγών και την απλοποίηση μετά το 2020. Κάναμε κάποιες αλλαγές και με το κανονισμό Omnibus που γνωρίζετε σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της κοινή γεωρικής πολιτικής. Βεβαίως, αυτό πάντοτε τίθεται υπό έλεγχο τη στιγμή το συζήτηση του PDP και δεν θα αλλάξει κάτι αυτή τη φορά. Όμως να ξέρουμε ότι η γεωργική πολιτική είναι η μόνη πολιτική που χρηματοδοτείται απόλυτα και είναι επιτυχής γιατί έχει παράξει παρκούς ποιότητας τρόφιμα για τους πολίτες, έχει βελτιώσει το κλίμα στις περιοχές της Πέδρου και έχει επίσης προσφέρει αξία στο ισοζύγιο πληρωμών. Ε, καθώς και στις εξαγωγές μας ε, έχουμε καταφέρει να ε, εξάγουμε προϊόντα καλής ποιότητας. Είναι επίσης σημαντικό για τους γεωργούς γιατί έχουν στήριξη στα εισοδήματά τους όχι μόνο για να επιβιώνουν, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στα εισοδήματα ε, των οικογενειών και στο μοντέλο των εκμεταλλεύσεων, αλλά έχουμε και έναν τομέα, μια ομάδα ανθρώπων που αποδίδουν όσον αφορά τα δημόσια αγαθά, δηλαδή το κοινό καλό, δηλαδή το κλίμα ε, ε, που αποτελεί όλο ένα και περισσότερο κομμάτι της πολιτικής ζωής, όπως επίσης ε, η προστασία των φυσικών πόρων. Θα δείτε αύριο στην ανακοίνωση για τη νέα κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2020 ότι θα υπάρχει απέτηση και προσδοκία όσον αφορά το υψηλό επίπεδο επίπεδο φιλοδοξίας για να μπορέσουμε να δούμε τις ε, συμφωνίες υψηλού επίπεδου ε, και στο πλαίσιο του, της διατροφής στο ΝΟΙΕ έχουμε ένα τομέα όπου πρέπει να κάνουμε περισσότερο σε σχέση με τα κοινά αγαθά και εφόσον αυτά χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των φορολογουμένων. Επίσης, για μετά την Brexit εποχή θεωρούμε πως θα έχουμε μια απώλεια σημαντική και βεβαίως θα πρέπει να βρούμε κάποια εξισορρόπηση στους ισολογισμούς μας. Εάν τα κρατημέλη της Ένωσης δεν θέλουν να συμβάλλουν επιπλέον πέρα από το 1% του ΕΠ, βεβαίως θα υπάρχουν περικοπές στις δαπάνες και στην γεωργία βεβαίως. Σε σχέση με το πρασίνισμα και την απόδοση αυτού, καθώς και το ποσοστό σφάλματος. Για την ετήσια έκθεση επιδόσεων για το 2016 έχουμε διαφορές γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα που ήταν αρκετά περίπλοκα και συμφωνώ πως πρέπει να τα ξαναδούμε και θα έρθω σε αυτό σε δύο λεπτά. Την πρώτη χρονιά όμως, το 2016, ήταν ε, περίοδος ε, εκμάθησης και για τους ε, γεωργούς. Δόθηκαν οδηγίες και βοήθεια. Είχαμε το σφάλμα για τις πληρωμές λίγο ψηλότερο, αλλά πάλι ήταν σε καλό επίπεδο και τα προγράμματα δράσης μας εφαρμόζονται για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Το ποσοστό σφάλματος λοιπόν ε, δεν έχει ε, αυξηθεί. Είμαστε στο 98% της εκτέλεσης. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν μέγα επίτευγμα και όπως είπα και νωρίτερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου χρειάζονται, χρειάζεται απλοποίηση και έχουμε διάφορα προγράμματα δράσης για την απλοποίηση που είναι υπό εξέλιξη. Τώρα, όσον αφορά την απόδοση του πρασινίσματος, 77% της γεωργικής μας γης είναι, καλύπτεται από κάποιο μέτρο πρασινίσματος και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, ωστόσο αποτελεί ένα, μια ένδειξη το, ότι το γεγονός ότι το 77% ο, της γης είναι υπό κάποιο πρόγραμμα πρασινίσματος και το 61,2% επίσης ε, ε, επηρεάζεται από ένα τουλάχιστον project. Έχουμε και τις ε, περιοχές οικολογικής εστίασης και αυτό είναι κάπως αντιφατικό κάποιες φορές, αλλά σαφώς έχουμε δείξει ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτή την πρόταση στη διάρκεια του έτους. Βεβαίως ε, υπάρχει ένα μια μεγάλη ζήτηση για πρωτεΐνη, έχουμε μέγα έλλειμμα και γι' αυτό και θα προτείνουμε στρατηγική πρωτεΐνης για το 2018. Θα συζητηθεί στις διάφορες επιτροπές εδώ, ε, ώστε να μειώσουμε την πρωτεΐνη που εισάγουμε από άλλα μέρη του κόσμου. Και ε, οι γεωργοί 14% έχουν επιλέξει ως ε, ε, περιοχές ε, οικολογικής εστίασης από την αρρώσιμη γη. Θέλουμε να μειώσουμε επίσης και το επίπεδο ζανικτώνων και παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις, σε αυτές τις περιοχές. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι η διαφοροποίηση της κοινή γεωρικής πολιτικής έχει, ε, έχει δυσκολίες στην εφαρμογή και πρέπει να περάσουμε και στην ε, μη ψησπορά. Ε, να έχουμε περισσότερη επικουρικότητα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε επίπεδο των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουμε ότι διατηρείται η κοινή γεωργική πολιτική που θα είναι στηριγμένη σε στόχου, σε επιδόσει, σε αποτελέσματα και όχι μόνο να βασίζεται σε κανόνε και κυρώσει. Φυσικά εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη αιρεσιμότητα σε σχέση με τα ε, χρήματα που δίνουμε στου γεωργού Αναφέρατε του νέου γεωργού στο κανονισμό Omnibus έχουμε ήδη συμφωνήσει για επιπλέον top-up στον πυλώνα 1 για τους νέους γεωργούς, 25% με 50%. Αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, ώστε οι νέοι να μπουν στη διαχείριση των, των εκμεταλλεύσεων, γιατί μόνο το 6% είναι νέοι κάτω των 40 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ε, πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, το 80% της γης ε, είναι η διοκτησία του 20% των γεωργών. Πρέπει όμως να δώσουμε επιλογές στα κρατημέλη, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Ορισμένες από τις επιλογές δεν έγιναν δεχτές όσον αφορά το κάπινγκ, την, το, πώς, τη φθήνουσα πορεία κτλ. Πρέπει να βρούμε περαιτέρω ιδέες και μέτρα. Με την πρόσφατη μας ανάλυση βλέπουμε ότι το 72% της βοήθειας που δίνεται στους γεωργούς ε, είναι αυτό που πάει στα 200 και 700 εκτάρια. Είναι σαφώς ε, ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Το 25% είναι αυτό των γεωργών. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει ανακατανομή στους μικρούς. Το κάπινγκ και σταδιακή μείωση θα πρέπει να γίνουν. Να αναφέρατε και την Αφρική, να πω με όλο το σεβασμό ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή και η γεωργική πολιτική επηρεάζει ε, και στρεβλώνει την αγορά στην Αφρική. Στην ε, διάσκεψη κορυφής του Ναϊρόμπι συμφωνήσαμε για την κατάργηση όλων των μεγάλων ε, επιδοτήσεων και ε, συμφώνησαν μαζί μας και είπα από την 1η του 2016 δεν υπάρχουν πια επιδοτήσεις στις εξαγωγές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αφρική ή στις άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου και αυτό είναι μέγα επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε βάλει στην ημερήσια διάταξη και ένα, και ένα έγγραφο θέσεων για την εγχώρια στήριξη. Ε, θα γίνει σχετική συζήτηση στον ΠΟΕ. Δεν ξέρω πώς θα τα πάμε εκεί, θα δούμε, αλλά δεν περιμένω και πολλά γιατί οι ΙΠΑ έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση στην συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς ε, έχουμε πολύ καλή συμμετοχή στην Αφρικανική Ήπειρο. Ε, και θα δούμε ότι η δική μας συμμετοχή θα φτάσει στα 440 δις ευρώ, όπως ανακοινώθηκε και από την εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να είναι επενδύσεις αυτά και συμφωνούσαμε και με την Αφρικανική Ένωση ότι θα υπάρχουν οδηγίες προς τις αφρικανικές χώρες αλλά και προς τις εταιρείες ε, της Ευρώπης ε, για το τι θεωρούμε υπεύθυνε ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον δηλαδή των επενδύσεων της ΕΤΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική. Και θα εξασφαλίσουμε δεν θα υπάρχει στρέβλος στην αγορά. Τώρα, Ρωσία και εμπάργκο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη στήριξή μας στους γεωργούς για τα οποροκυπευτικά τα τελευταία χρόνια αυτό είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα για πολλούς από τους γεωργούς μας γιατί δεν καταφέραν να αντικαταστήσουν ε, ε, την αγορά που είχαν με τις εξαγωγές προς τη Ρωσία. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί οι τομείς, ε, ο τομέας των απορροκυπευτικών δεν το κατάφερε αυτό ενώ το καταφέραμε σε άλλους τομείς τροφίμων. Πρέπει μέχρι του χρόνου να το καταφέρουμε ε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και το πρόβλημα του ρωσικού εμπάργου. Ρωτήσατε για το ειδικό ζήτημα της Τσεχίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Εμείς ξεκινήσαμε διαδικασία μέσα στο 2016 όσον αφορά την ε, παραβίαση των κριτηρίων ε, του οργανισμού πληρωμών. Πρόκειται για κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί από την νομοθεσία και η διαδικασία συμμόρφωσης συνεχίζεται. Σεβόμαστε τις ε, προθεσμίες και έτσι δεν μπορώ να το σχολιάσω πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Ελπίζω να απάντησα στις ερώτησεις σας. Ίσως η τελευταία ερώτηση ήταν ο ορισμός του Γεωργού σύμφωνα με την, τον κανονισμό Omnibus Bad, ε, με τον κανονισμό του Omnibus είπαμε θα ισχύσει περισσότερη επικουρικότητα και ότι τα κράτη-μέλη θα ορίσουν τι είναι ο ενεργός ε, γεωργός ε, τελικά όμως στάσαμε σε έναν κατάλογο αρνητικών δηλώσεων για το τι δεν είναι ένας δραστήριος ε, ή ενεργός γεωργός. Θα έπρεπε δηλαδή κατά τη γνώμη μου αυτός να ασχολείται με την ίδια τη γεωργία και όχι απλά με επενδύσεις. Αυτά και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και για μας, για την Επιτροπή μας δηλαδή, τι είστε το ερώτημα ε, τι γίνεται στην Αφρική λόγω των ευρωπαϊκών πλεονασμάτων αλλά και των πληρωμών, των αμέσων ενισχύσεων. Είναι σημαντικό θέμα και για μας, ας πούμε στη Γερμανία. Δεν υπάρχει αναφορά στην τηλεόραση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που να μην μας προσάπτει ότι έχει κλείσει ένα εργοστάσιο στην Αφρική ή γυναίκες που δεν μπορούν να πουλήσουν στα παζάρια τα προϊόντα τους γιατί τους έχουν κατακλείσει οι ευρωπαϊκές εισαγωγές. Και ποδαβλίζεται έτσι ένα αντιευρωπαϊκό αίσθημα στον πληθυσμό και ε, κυριαρχεί από τη μια αυτό. Από την άλλη μας έρχονται πρόσφυγες γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν στην Αφρική. Τι είστε το ερώτημα. Ε, ποια είναι η σχέση των δικών μας πολιτικών με άλλα μέρη του κόσμου και τι αποτελέσματα έχουν. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Σκιώδης συζητητές, η κυρία Γιάλα Σέντερ πρώτη, παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Πίτρο Πεχόγκαν. Για να είμαι ειλικρινή, όπως έγινε και χθε με την κυρία Τέισεν, οι προτάσεις και οι ερωτήσεις μας και του κυρίου Τσέλερ ε, μας έχουν καλύψει γιατί ήταν πάρα πολύ πλήρης η αναφορά του εισήγητου. Απλώς εγώ θέλω να σας κάνω κάποιες μικρές ερωτήσεις, πιο πολύ ανησυχίες να σας μεταφέρω. Εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από το καθένα, γιατί αύριο αρχίζει να λασάρετε αυτή την ανακοίνωση για το μέλλον. Η απαλλαγή του 2016 συμπίπτει με σημαντικές αποφάσεις παράλληλα για το Brexit και για την αρχική πρόταση του κυρίου Τίνκερ για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο και δεν σας κρύβω ότι έχει αρχίσει εδώ και κυκλοφορεί η φήμη ότι θα πληρώσει την ύφη η κοινή γεωργική πολιτική αν δεν βρούμε κανένα άλλο εξελαστήριο θύμα. Εγώ ως Ισπανίδα δεν συμφωνώ προφανώς με αυτό καθόλου και ακριβώ αν χρειαστούν θυσίες θα πρέπει αυτές να μοιραστούν στις διάφορες πολιτικές και να μην την πληρώσει η γεωργία. Υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τις ενισχύσεις και πώς θα επηρεάσουν την ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες. Μεσογειακές. Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες εγκαθίστανται ε, ε, και στην νότια όχθη της Μεσογείου και βοηθούν εκεί για την ανάπτυξη της γεωργίας αυτά τα κράτη. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί ε, και εργασία δίνουν και αναπτύσσουν και βελτιώνουν τη γεωργία των κρατών αυτών. Κάποια στιγμή χρειάζεται κάποια εξορρόπηση. Παρ' όλα αυτά ανησυχώ όμως, ανησυχώ όπως σας είπα, γιατί κυκλοφορεί αυτή η φήμη ότι θα κάνετε περικοπές. Εσείς πώς το σκέφτεστε, πώς θα θέλετε να ενισχύσετε την επιχειρηματολογία και στις άμεσες ενισχύσεις αλλά και στην αγροτική ανάπτυξη που είναι πιο δύσκολο γιατί ήταν πολύ πιο περίπλοκες οι διαδικασίες με συνυπευθυνότητα, συγχρηματοδότηση και υπάρχουν και αρνητικές πτυχές με τα σφάλματα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρατε και μπράβο σας. Ε, υπάρχει σημαντική βελτίωση. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνω, επειδή στο μέλλον έχουμε τα προβλήματα που είπατε, υπερβολική ευελιξία στα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν κάποια πρότυπα, κάποιοι κανόνες που προσπαθούμε να ανταποκρίνονται σε στόχους και σε αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση που ελήφθη το 2013 να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη έχουμε μια αναντιστοιχία από τη μια εμείς απαιτούμε να έχουμε αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένους στόχους, τα γνωρίζετε αυτά και με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη και ελευθερία κινήσεων, οπότε ορισμένα μέτρα χωλένουν. Όπως είπατε και εσείς, ο ορισμός του ενεργού αγρότη, η συμμετοχή των νέων αγροτών στη χώρα μου. Είναι πολύ περίπλοκο και πολύ δύσκολο. Αύριο λοιπόν στην ανακοίνωση που θα παρουσιάσετε Ποια είναι τα μέτρα εκείνα που θα σας επιτρέψουν να εξασφαλίσετε τα κράτη-μέλη να μας βοηθήσουν, να βοηθήσουν τον εαυτό τους τον ίδιο για να προχωρήσουμε ε, στη μελλοντική πρόταση. έτσι ώστε η ΚΑΠ μετά το 2020 να είναι πιο κοντά στο πρασίνισμα, ε, στην ε, ένταξη των νέων αγροτών, στη βελτίωση της γεωργικής δραστηριότητας και όλα αυτά που έχουμε ως στόχους. Καινοτομία, πρόοδος και πώς θα περιορίσουμε αυτή τη χαλάρωση των κρατών μελών που προκαλεί προβλήματα είτε για λόγους συγχρηματοδότησης είτε για άλλους διαδικασιών. Επίσης, μιλάτε για πρασίνισμα, για πρόθεση της οικολογίας, για μείωση των φυτοφαρμάκων και των ζυζανιοκτώνων. Αλλά βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πάρα πολύ ε, και πάρα πολύ γρήγορα τη γεωργία, πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Τη γεωργία όχι μόνο του Νότου αλλά και του Βορρά. Προβλήματα βλέπουμε και ε, αλλού. Όλο και πιο νωρίς ε, έχουμε τον τρίγο στις χώρες του Νότου και ε, βλέπουμε επίσης και πιο βόρειες χώρες για λόγω της κλιματικής αλλαγής να καλλιεργούν αμπέλια, όπως είναι το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία. Ε, υπάρχουν προβλήματα από τη λειψιδρία επίσης και την ξηρασία για τους αγρότες. Ε, εσείς σκοπεύετε να βοηθήσετε για να αντισταθμιστούν αυτές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έχετε προβλέψει από τώρα τα μέτρα για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων περιορισμών και των θεομηνιών που αναμένονται και φαίνονται ήδη δηλαδή λόγω των κλιματικών αλλαγών. Επίτροπος παρακαλώ. Α, κύριε Επίτροπε, έχουμε άλλους επτά συναδέλφους για να το έχετε υπόψη σας έτσι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γιαλασέντερ. Συμφωνώ με το αίσθημα της κυρίας Αγέλα Σέντερ για το μέλλον της ΚΑΠ, τις ευαισθησίες, τις ευθύνε, πώς μπορούμε να τις επιμεριστούμε μεταξύ κρατών μέλων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επιτυχής αρκετά σε θέματα ανταγωνισμού. Προσέθεσε τεράστια αξία διασυνοριακά. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλους. Αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών και των 28. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε έναν τρόπο να αποκτήσουν περισσότερη λογοδοσία τα κράτη-μέλη για τους στόχους που θέτουμε βάσει δικτών, στόχων στο πλαίσιο των πολιτικών μας αυτή τη στιγμή Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν σε ιδιαίτερες συνθήκες. Πώς μπορεί η ΚΑΠ ε, να επιτελέσει ε, τα όσα της ανατίθενται. Ε, οι συνομοθέτες θα τα αποφασίσουν, δεν κάνω μόνο εγώ προτάσεις και εσείς θα έχετε να πείτε μια άποψη για το τελικό αποτέλεσμα, για το τι θα γίνει η ΚΑΠ. Έχετε δίκιο. Δεν θα είναι εύκολο ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον προπολογισμό και δεδομένου του Brexit θα αλλάξουν πολλά πράγματα και μετά έχουμε και τις περισσότερες δαπάνες σε διάφορα θέματα όπως η ασφάλεια, η προστασία των συνόρων, μετανάστευση. Οπότε στο μέλλον ε, θα αλλάξουν τα πράγματα. Σε σχέση με τους νέους αγρότες, είναι θέμα επιμερισμένης διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει παραπεριορισμένα πράγματα γιατί στα θέματα ε, φορολογίας ε, είναι αρμόδια τα κρατη Και κάποια κάνουν ε, σωστή δουλειά, αλλά χρειάζονται να γίνουν περισσότερα για να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες, να εμπλέκονται περισσότερο στο διαχειριστικό κομμάτι των αγροκτημάτων από ότι τώρα. Να τους δώσουμε κίνητρα μέσω ευρωπαϊκών μέσων και ενδεχομένω και χρηματοδοτικών μέσων όταν σε κάποια κράτη-μέλη είναι δύσκολο να γίνουν κεφαλακές επενδύσεις ε, όταν αναλαμβάνει ένα αγρόκτημα κάποιο νέος άνθρωπος. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα χρηματοδοτικό μέσο για να βοηθήσουμε τους νέους να, εμπλακεί, να εμπλακούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, είτε εξ αρχής είτε μετά από κληρονομιά. Το πρασίνισμα που αναφέρατε, οι σχετικές πρακτικές ε, έτσι όπως υλοποιούνται είναι ε, περίπλοκες βάσει των ανησυχιών που εκφράζουν οι γεωργοί. Παρ' όλα αυτά στις αιτήσει ε, για πληρωμές που κάνουν οι γεωργοί ε, η νομοθεσία απαιτεί 5% περιοχές οικολογικής εστίασης και αυτοί αιτούνται 14%. Οπότε είτε αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν τις συνολικές νομοθετικές απαιτήσεις και περνάνε το όριο, κατά πολύ το αναμενόμενο όριο που αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση ε, φοβούνται δηλαδή για το χαρακτηρισμό διαφόρων περιοχών των ε, χέρσων γεών των... το 77% των συνολικών αρρώσιμων περιοχών υποκείται σε απαιτήσει ε, διαφοροποίησης και υπόκειται σε EFA αλλά το 14% έχει δηλωθεί ως EFA αυτό είναι ένα ε, επίμαχο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Για τους μόνιμους λιμόνες, 29% ε, αποτελούν τη συνολική ε, αρρώσιμης περιοχής και σε κάποιες χώρες είναι το 90% από το οποίο μεγάλο κομμάτι είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Και μετά αυτό που αναφέρεται για τις φυσικές καταστροφές, οι πυρκαγιές στην Ισπανία, στην Πορτογαλία για παράδειγμα, οι πλημμύρες ε, Στι χώρε τη Βαλτική, στη Φιλανδία, αποτέλεσαν σημαντικά ζητήματα για διάφορους λόγους ε, στη Μεσόγειο και στην Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη. Πρέπει να αναζητήσουμε να βρούμε μέτρα καταλληλότερα για την διαχείριση των κινδύνων προς όφελος των αγροτών αλλά και των ε, αγροτικών κοινοτήτων. Η ευελιξία που δείχνουμε στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για προπληρωμές ή για επαναπρογραμματισμό για αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών λειτουργήσαν πολύ καλά το 2017. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα στο πλαίσιο της κλιματικής δράσης που μπορούμε να υιοθετήσουμε αναγνωρίζοντας ότι το κλίμα είναι σημαντικός παράγον για το μέλλον και που θα πρέπει να ε, ε, ληφθεί υπόψη στην πολιτική μετά του 2020. Η κυρία Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που απαντήσατε σε όλες μας τις ερωτήσεις. Κάθε χρόνο έχουμε όλο ένα και πιο πολλές ερωτήσεις και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά είναι πολύ καλή αυτή η πρακτική και για μας και για την Επιτροπή πιστεύω. Έχω μια ερώτηση μόνο γιατί την υπέβαλα και χτες στην Επίτροπο Τάισιν και μάθαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά το ή ελάχιστα σε σχέση με το σχέδιο για το απλοποιημένο κόστος. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε αποτελέσματα για τη χρήση αυτού και όλοι γνωρίζουμε ότι το απλοποιημένο κόστος περιορίζει το διοικητικό φόρτο των δικαιούχων και το κίνδυνο σφάλματος γιατί χρειάζεται να προωθηθεί η χρήση του απλοποιημένου κόστους ο κανονισμός 1307 ε, διευκολύνει τους μικρούς γεωργούς, αλλά ορισμένα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν. Γι' αυτό ρωτώ εσάς και το ελεκτικό συνέδριο, γιατί κάποια κράτη-μέλη διστάζουν τόσο πολύ και είναι απρόθυμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το, το σχέδιο απλοποιημένου κόστους και πόσο επιτυχώς έχει προωθήσει η Κομισιόν αυτό το project για να μειωθεί το διοικητικό κόστος και ε, το σφάλμα. Θα το αναπτύξετε περαιτέρω, καθώς προχωράμε μετά το 2020 και το νέο PDP και το νέο κανονισμό ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πώς θα το κάνετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε ε, την πραγματική απλοποίηση μέσω αυτού του προηγουμένου κόστους και επίσης μήπως μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την αυριανή ανακοίνωση γιατί αν δεν το μοιραστείτε με την αγαπημένη σας Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, με ποιον θα το μοιραστείτε αυτό το την καινούργια ανακοίνωση. Κύριε Επίτροπε, ορίστε αφού σας ρωτάει και τέτοια πράγματα η συνάδελφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καμπάγιουβα. Για το απλοποιημένο κόστος και τη σχετική επιλογή και εγώ είμαι υπέρ. Όπω και εσεί, έχουμε κάνει κάποιε αλλαγέ στο Omnibus για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτέ τι επιλογέ κόστου ορισμένα συγκεκριμένα εμπόδια έχουν αφαιρεθεί από τη Συμφωνία Omnibus και ε, δεν περιλαμβάνεται ο, η μέθοδος υπολογισμού όσον αφορά την το απλοποιημένο κόστος. Αντίθετα, ε, ο υπολογισμός ε, λαμβάνεται υπόψη αργότερα και αυτό είναι σύμφωνο με τα υπόλοιπα τα κονδύλια ε, των Ταμείων της Ένωσης. Ελπίζομαι ότι θα βρεθεί συμφωνία σύντομα και η Επίτροπος Τάισεν κάνει μεγάλη προσπάθεια, συνεργαζόμαστε στενά ώστε να αναπτύξουμε ε, κοινού κανόνες. Δεν είμαι σε θέση να μοιραστώ μαζί σας περισσότερα για την ανακοίνωση στην Αυριανή. Επιτρέψατε μου να τα ε, <laughs> πω αύριο, αλλά Είμαι βέβαιος ότι του χρόνου θα έχετε την ευκαιρία να με ρωτήσετε τι κάνω για όλα αυτά που θα ανακοινώσω αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάναγκαν παρακαλώ. Ευχαριστώ. πολύ. Σε σχέση με τα ποσοστά ασφάλματος, ε, το επαναλαμβάνω διαρκώς, τα πραγματικά ασφάλματα Κάποιοι προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν ως απάτες, αλλά είναι πραγματικά ασφάλματα. Ξέρετε, το ασφάλμα είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν μπορεί κανείς ε, ως άνθρωπος να καταλάβει την περιπλοκότητα όλων αυτών των συστημάτων. Ε, ελπίζω ο κ. Χόγκαν να έχει μια καλή ανακοίνωση για μας αύριο, διότι όπως φαίνεται ο πυλώνας 1 ε, έχει προτεραιότητα όσον αφορά την απλούστευση. Αλλά οι φτωχότεροι αγρότες ε, του πυλώνα 2 δεν καταλαβαίνουν τα πράγματα σε βαθμό που πολλοί κόσμος έρχεται σε εμά με τόσες πολλές απορίες ε, ε, ξανά και ξανά όπου κάνουν σφάλματα, οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν κάνει σφάλματα, ενώ αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των συστημάτων. Και σε πολλές περιπτώσεις στέλνουμε ε, Ενημερώσει ε, για το πώ λειτουργούν τα συστήματα και μέχρι αυτό να πάει στους αγρότες έχει αλλάξει διατύπωση και αυτό γίνεται ξανά και ξανά και η Κομισιόν λέει «Α, είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους». Και, και ξέρετε αυτό δεν είναι μία περίπτωση, φαίνεται να γίνεται διαρκώς. Είναι συστημικό το θέμα. Τι θα κάνει η Κομισιόν γι' αυτό, διότι οι αγρότες θέλουν να ε, ακολουθήσουν το σύστημα αυτό, αλλά είναι αδύνατον η Κομισιόν μάλιστα ζήτησε από έναν αγρότη να μιλήσει σε σύμβουλο. Είναι τα συστήματα τόσο περίπλοκα και εγώ ήμουν σύμβουλος μέχρι πριν από δύο εβδομάδες και εγώ πάλι δεν καταλάβανα. Όταν μιλάμε για ασφάλματα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των συστημάτων. Αυτό πρέπει να αλλάξει μου κάνει εντύπωση όταν ακούω κάποιον από τελείω ε, άλλη πολιτική ομάδα, από τη δική μου, τον κύριο Τσέλερ, να μάχεται διαρκώ για να αλλάξει την κατάσταση, όπου το 80% των χρημάτων πάει στο 20% των αγροτών. Έχω να σα πω κάτι ενδιαφέρον, κύριε Τσέλερ. Στην Ιρλανδία, αν έρθετε, θα σα πούνε ότι είστε κομμουνιστή. Αυτό είπαμε και εμεί στι τελευταίε διαπραγματεύσει ε, για την ΚΑΠΑ, Το είπε ο Τζον Μπράιν από το μεγαλύτερο οργανισμό γεωργών. Μίλησε για σύγκληση, για ισότητα, για ε, προοδευτική μείωση ε, ως κομμουνιστικές ιδέες. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Με αυτόν έχετε να κάνετε. Αυτός ο άνθρωπος ε, ο οποίος ανέφερε αυτό που προτείνετε και εσείς ως κομμουνισμό κατέστησε το Χόγκαν στη Βουλή και έτσι έχουν... Δεν χρειάζεται να απαντήσω τελευταίο ε, κομμάτι, είναι γνώμη του κ. Φλάναγκαν. Ο κ. Τσέλερ θα αποφασίσει αν θέλει να μας πει αν είναι κομμουνιστής ή όχι. Αλλά σε σχέση με τις αλλαγές και τα σφάλματα και τις απάτες, προφανώς η απάτη και το σφάλμα δεν είναι το ίδιο. Όταν μιλάμε για σφάλματα, για ποσοστά τον ε, εννοούμε σφάλματα και όχι απάτες και από τη συζήτηση σήμερα φαίνεται ότι έχουμε ένα ε, στιβαρό ε, σύστημα διαχείρισης ε, στην έκθεση του 2016 της Όλαφ. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσει απάτη σε θέματα ΚΑΠ. Οι παρατυπίες την τελευταία πενταετία αντιστοιχούν μόλι στο 0,001%. Ελάχιστο κλάσμα αυτού για το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Αγροτικών Εγγύσεων. Είναι πολύ χαμηλό πιστεύω το ποσοστό. Όσον αφορά την απλούστευση τη πολιτική, συμφωνώ με τον κύριο Φλάνναγκαν, Πρέπει να κάνουμε πολλά ε, περισσότερα. Είναι επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε τα συστήματα ε, και αξιοποιούμε καλά τα χρήματα των φορολογουμένων για να βοηθήσουμε τους αγρότες Τώρα, όσον αφορά τι ενισχύσει του πυλώνα 1 και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι γεωργοί όσον αφορά τι αιτήσει του για βασικέ ενισχύσει, έχουμε κάνει σημαντικέ αλλαγέ την τελευταία διετία και απλούστευση. Τώρα έχουμε έναν προληπτικό ε, έλεγχο που εξελίφθη τα μικρά ασφάλματα που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα και από πολιτική άποψη ε, σε πολλούς ε, από τους γεωργούς μας διότι μπορούσαν να χάσουν όλες τους ενισχύσεις για ένα πολύ μικρό σφάλμα. Αυτό ήταν άδικο. Οπότε έχουμε εισάγει και ένα σύστημα ε, κίτρινης κάρτας που σημαίνει ότι αν αποδειχθεί ότι το σφάλμα είναι γνήσιο στα κράτη-μέλη τους δίνουμε μια αναλογική μείωση ε, διοικητικών ε, ποινών αλλά και κάποιο περιθώριο να διορθώσουν τα ασφάλματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, έχουμε μια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινή λογική. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να έχουμε και συστήματα προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Δηλαδή αυτή η ισορροπία πιστεύω μεταξύ απάτη και πραγματικών σφαλμάτων έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπω βλέπετε και από τα νούμερα που σα έχω δίνει, τα περισσότερα σφάλματα, mm. τα σφάλματα που εμεί αναγνωρίζουμε είναι πραγματικά σφάλματα και όχι απάτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Καλωσορίσατε, μάλιστα στην Επιτροπή μας. Ήθελα να πω ότι ποσοστό σφάλματος 2,5% είναι πολύ ικανοποιητικό δεδομένου του παρελθόντος. Ε, τώρα δεύτερον, δεδομένης της σύγχυσης που προκάλεσαν όλα τα στοιχεία πρασινίσματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν πάει πάρα πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε θέλω να συγχαρώ τον Επιτροπό και όλου του ε, εμπλεκόμενου. Θεωρώ ότι όλα αυτά δείχνουν ότι το σύστημα την χάνει σωστή διαχείριση και ότι κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε προτείνω να συνεχίσουμε προ την ίδια κατεύθυνση και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω απλούστευση. Ωστόσο, συμφωνώ, θα υπάρξουν νέε προκλήσει για το σύστημα ανεξάρτητα του Brexit, ακόμη και αν δεν γινόταν το Brexit, είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση του τομέα μέσω ποσοστού των συναλλικών δαπανών της ΚΑΠ έπρεπε να μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε στόχους στο μέλλον. Πέραν της προσθέμενης αξίας θα πρέπει να εστιαστούμε όλο και περισσότερο στα αποτελέσματα του τομέα. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Ένα από τα διαρκή προβλήματα είναι η διάκριση μεταξύ όσων ασχολούνται με τη διαχείριση υγιής και την παραγωγή τροφίμων ε, και μεταξύ των συμφερόντων ε, όσων ασχολούνται με την γεωκτησία ε, και τη... αυτό υπήρξε ανέκαθεν ένα μεγάλο ζήτημα και αποτελεί όλο και μεγαλύτερο χάσμα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ όσων κατέχουν τη γη και όσων ε, την δουλεύουν ε, ενεργά. Τα συμφέροντα τους δεν συμφωνούν πάντα. Οπότε προτείνω η επανεστίαση στα αποτελέσματα να σημάνει ε, νέες προσπάθειες υποστήριξη. Ευχαριστώ. Well, I can summarize my Ωραία, θα συνοψίσω την απάντησή μου με τον κύριο Ashworth, στον κύριο Ashworth λέγοντας ότι συμφωνώ με τόσα λέει. Μας εκπλήσει πρέπει να πω ότι το ποσοστό σφάλματο ε, για το πρασίνισμα είναι τόσο χαμηλό. Διότι όταν εισήγαμε αυτό το σύστημα το 2013 και το θεώρησαν οι γεωργοί μα και τα κράτη-μέλη μα τόσο περίπλοκο, καταλαβαίνετε ότι μα εκπλήσει και εμά και το ελεκτικό συνέδριο ότι είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό σφάλματος. Οπότε πρέπει να συγχαρούμε του ανθρώπου που ανεπλάξαν στη διαδικασία ε, και την εφάρμοσαν τόσο καλά με τις σωστές, δεν σωστέ σωστές οδηγίες ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Οπότε συμφωνώ μαζί σας. Συγχαίρω και εγώ το προσωπικό μου στην DJ Agri και τα, στα κράτη-μέλη ε, που τα κατάφεραν τόσο καλά στην υλοποίηση αλλά χρειάστηκε πολύ χρόνο το 2015 ε, για την υλοποίηση αλλά απέφερε αποτελέσματα ε, πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στα αποτελέσματα παρά να έχουμε μια προσέγγιση επικεντρωμένη σε κυρώσεις κάτι που δημιούργησε προβλήματα σε ανθρώπους σε πολλές χώρες ο ορισμό του ενεργού αγρότη, όπω γνωρίζετε από την τελευταία μεταρρύθμιση, είναι δύσκολο. Οπότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε να υποστηρίζουμε του ενεργού γεωργού, αυτού που σηκώνται νωρί το πρωί και δουλεύουν τα αγροκτήματα για να ζήσουν τι οικογένειέ του. Ο γεωργικός τομέας είναι αυτό που είναι η Καθολική Εκκλησία ε, παγκοσμίω. Κα, κανείς ε, δεν έχει τόση εμπειρία συγκεντρωμένη όσο εσεί. Αν δεν τα καταφέρετε εσεί, ποιο θα τα καταφέρει. Ε, ο κύριο Αλαφράνκα, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τι εξηγήσει που μα δώσατε. Προφανώ η κοινή γεωργική πολιτική είναι μια πολιτική που γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχε ως στόχο να εγγυηθεί ένα εισόδημα στους αγρότες μας, αλλά και να έχει ευρωπαϊκή αγορά σωστά γεωργικά προϊόντα με καλή διανομή. Και η πολιτική αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, είναι σαφές. Πλην όμως άλλαξαν οι συνθήκες και το περιβάλλον, οπότε γι' αυτό χρειάζεται ε, να μεταρρυθμιστεί η πολιτική αυτή. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Τσέλερ, το εξήγησε πολύ καλά. Απορροφά 40% του ευρωπαϊκού προπολογισμού η πολιτική αυτή. Και προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η δαπάνη, αλλά και η δαπάνη που να πιάνει τόπο και να φτάνουμε στους στόχους μας. Και χαιρόμαστε που έχει μειωθεί και το ποσοστό σφάλματος. Θα ήθελα να σας πω κύριε Επιτροπέ ότι με ανησυχεί η κατάσταση των νέων αγροτών μας εκεί αφιερώνουμε σημαντικούς πόρους και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι φτάνουμε στους επιθυμητικούς στόχους. Έχετε δίκιο που αναφερθήκατε ε, ε, στα πρότυπα ε, που αναπόκειται στα κράτη-μέλη να ορίσουν πώς θα γίνεται η διαδοχή σε μία εκμετάλλευση. Έχετε στοιχεία για το πώς είναι οι νέοι αγρότες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό του ενεργού πληθυσμού. Είναι πολύ βασικά στοιχεία. Ο αγροτικός πληθυσμός ε, σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο είναι και πόσο είναι η συνεισφορά της γεωργίας διακόπτη μιλητής κατά πόσο λοιπόν συνεισφέρει η γεωργία στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Τσέλερ για τα σφάλματα που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά ε, τις επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι οι οργανισμοί πληρωμής δεν έχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις ε, χρήσεις γης, για τις κατηγορίες γης, για τις άμεσες ενισχύσεις. Το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης επίσης έχει σφάλματα σε σχέση με κάποιες γης που δεν δικαιούνται επιδότηση και επίσης αυτά τα σφάλματα ε, για δικαιούχους που δεν είχαν αποκαλύψει όπως ε, επιβάλλουν ευρωπαϊκοί κανόνες ή εθνικοί κανόνες τη σχέση τους με τις εταιρείε που ελέγχουν ε, τις καλλιέργειες. Και τέλος, για ε, τις εκθέσεις Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπάρχουν ανεπάρκειες σε εκθέσεις και ζήτησε να βελτιωθούν οι δειγματοληψίες, τα, τα δείγματα και οι υπολογισμοί των επιπέδων σφάλματος. Χαίρομαι κύριε Επίτροπε που λαμβάνετε σοβαρά υπόψη ε, τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και που θα μελετήσετε πώς θα βελτιώσετε αυτές τις ελλείψεις ή τις ε, ασάφειες. Μια τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε, για να μην μακρηγορήσω. Στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο έχουμε μια νέα εμπορική πολιτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την έλευση του ε, νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θετικό ισοζύγιο και εμπορικό, αλλά και ε, ισοζύγιο αγαθών, ε, γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κύριε Επιτροπέ, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Θα πρέπει να βρούμε κάποια μορφή ισορροπίας ανάμεσα στις αρχές που διέπουν ε, το μοντέλο μας του ελεύθερου ανταγωνισμού σεβόμενοι πάντα τους κανόνες που ε, διέπουν τη συμμετοχή σε μία λέσχη ας πούμε που είναι η ευρωπαϊκή και η γεωργική πολιτική. Το νέο αυτό εμπόριο δεν ε, σημαίνει μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ σκέφτεστε μέτρα για να ανακουφιστούν ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι εμπορικές μας συμφωνίες και πώς θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνουν ε, ενδεχομένως κάποιες νέες αγορές που ανοίγουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα Σάντσες για τους νέους ε, γεωργούς. Συμμερίζομαι την ανησυχία σας ε, για τους νέους και την ανάγκη να προσελκυστούν νέοι άνθρωποι στη Γεωργία. 6% του πληθυσμού μας ε, στη Γεωργία είναι κάτω των 40 ετών. Δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση όσον αφορά την μελλοντική ανταγωνιστική Γεωργία. Στη μεταρρύθμιση του 2013 εισήχθη η η στήριξη στους νέους ε, για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους και από το 25% πήγε στο 50% μέσω του Omnibus. Το 2016 σχεδόν 20.000 ε, νέοι ε, πήραν αυτή την άμεση πληρωμή, πήραν συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ. 177.000 νέοι ε, είναι προγραμματισμένοι να λάβουν, να λάβουν βοήθεια στην περίοδο 2014 με 20 και έχουμε και επιπλέον στόχους μέτρησης αλλά και επιδότησης ε, μέσω του προγράμματος ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτά είναι γενικά τα μέτρα που λαμβάνουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικά. Αρκετά αποτελεσματικά, μάλλον όχι από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και μοιραζόμαστε με τα κράτη-μέλη τι δικές τους δράσει όσον αφορά τη φορολόγηση. Αυτό είναι στη δική τους ε, αρμοδιότητα. Αλλαγέ στη φορολογία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα είναι θέμα κλειδί. Αλλά θα δείτε και ότι ε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο για να προωθήσουμε ε, τους νέους στην Γεωργία. Για σε περιοχές οικολογικής ε, εστίασης είχαμε ένα στόχο 5% αλλά η εφαρμογή όπως είπα νωρίτερα έχει οδηγήσει το 14% ε, να καλύπτονται ε, από αυτό το μέτρο της οικολογικής εστίασης το οποίο στόχος ήταν να βοηθήσει τη βιοπικιλότητα. Δεν ξέρουμε αν είχε μεγάλο αντίκτυπο μετά από ένα χρόνο, είναι κάπως νωρίς. Αλλά, ε, ωστόσο, οι γεωργοί ανταποκρίνονται. Υπήρξαν κάποιες απόψεις από τους γεωργούς ότι πρόκειται για μια, ένα απότομο, ένα ομό μέσο, να εντοπίσουμε δηλαδή ένα κομμάτι γης ε, ως ε, ε, σύνορο ή ως ζώνη ανακοπής, αναχέτησης πάντως ενδιαφέρονται να το κάνουν ε, επειδή ε, ε, λαμβάνουν την οικονομική στήριξη. Όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα γιατί τα δημόσια αγαθά είναι σημαντικά. Το κοινό καλό είναι σημαντικό και οι γεωργοί φαίνεται να είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν εδώ και αύριο θα πω περισσότερα γι' αυτό επίσης. Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν φοβούμε καθόλου τις εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε συνάψει πολλές τα τελευταία χρόνια με το Βιετνάμ, με την Ιαπωνία, με τη Σιγκαπούρη που πρέπει να κυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και τη ε, κράτη-μέλη, τον Καναδά βεβαίω, και αναμένουμε να επιτύχουμε και τα συμπεράσματά μας με το Μεξικό και Μερκοσούρ. Αλλά είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει για τα όσα είπατε. Ε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο τι μπορούμε να παζαρέψουμε στου διαφορου τομεί προ όφελο, συνολικά τη Ένωση και όλων των τομέων. Και η Γεωργία πιέζεται σε μια διαπραγμάτευση με το Μερκοσούρο που είμαστε αμυντικοί σε σχέση με όλα σχεδόν. Και έχουμε αυτό το κλασικό δίλημα όπου ίσως ο γεωρικός τομέας ανησυχεί για ολόκληρη την οικονομία και πρέπει να μπορέσουμε να, βρούμε μια ισορροπία, να βρείτε μια ισορροπία γενικά για το καλό ολόκληρη της Ισπανίας. Τέτοιου είδους προκλήσεις αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Και Βεβαίω προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουμε ισορροπημένη συμφωνία για ευκαιρίε επιθετικέ και αμυντικέ. Σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Και αυτό κάνουμε σε όλε τι συμφωνίε που πρέπει να συναυθούν. Και έχουμε και θετική, θετικό ισοζύγιο με την Ιαπωνία. Πιεζόμαστε λίγο για το Μερκοσούρ, αλλά ελπίζω ότι αν έχουμε μετριοπαθεί προσδοκίε μπορούμε να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία που δεν θα απαιτηθεί αυτό το είδους το ταμείο το οποίο αναφέρατε στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σαβαρμά και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον ε, πρόεδρο της Πετροπολής Γεωργίας, τον κύριο Σικέσκι. Thank you, Chair. Ο κύριος Σαβαρμά, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χόγκα, κύριε Επίτροπε και τον εισηγητή μας βεβαίως. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε στη σημερινή συζήτηση. Δεν περιμένω να λάβω συγκεκριμένη απάντηση, αλλά κάτι με βασανίζει. Αν έχουμε συλλέξει ε, ε, τις σωστές πληροφορίες από αυτά που ακούμε που θα ανακοινώσετε αύριο και από τα όσα μας λέτε εδώ σήμερα, κύριε Επίτροπε, Στην επόμενη κοινή γεωργική πολιτική θα υπάρξει μετατόπιση προς μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα διάφορα προγράμματα και συστήματα και ταυτόχρονα θα δοθεί πολύ περισσότερη έμφαση, ακόμα πιο πολύ, στο πρασίνισμα. Όπως γνωρίζουμε, σε ορισμένα κράτη-μέλη, λοιπόν, Ο λόγος των Βρυξελών είναι Ευαγγέλιο. Και υπάρχει μια τάση να έχουν ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι οι Βρυξέλλες, που μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Διερωτώ με λοιπόν, α, και βάζω και ένα τρίτο στοιχείο εδώ, την απλούστευση, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να την κουβεντιάζουμε και περιμένουμε κάτι να γίνει, κάτι περισσότερο. Πολλοί να έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα υπό τη δική σας ηγεσία, κύριε Επίτροπε, με την τελευταία διετία. Αλλά τι θα συμβεί. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ερώτηση και με ενδιαφέρει να ακούσω την απάντησή σας. Τι θα συμβεί μετά το 2020 όταν τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και όταν έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποιο κοινή γεωργική πολιτική. Φοβούμε ότι θα καταλήξουμε μάλλον σε μια συγκεχημένη κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη. όπου αν υπάρξει ευελιξία, η οποία είναι καλή και άγια και σπουδαία ιδέα, δεν διαφωνώ, αλλά πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να φροντίζει ότι θα έχει κάποια συνοχή η πολιτική αφενός και αφετέρου δεν θα έχουμε ακόμα πιο περίπλοκες διαδικασίες, συστήματα που οδηγούν σε σύγχυση στα κράτη-μέλη, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει και σε ένα ακόμα στρώμα ε, διατάξεων, ας πούμε, και γραφειοκρατίας μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτο. Αν καταλαβαίνετε αυτό που προσπαθώ να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ε, τα βρω όλα αυτά που ρωτάτε φυσικά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Όλοι λένε ότι η πολιτική είναι πολύ περίπλοκη. Οι αγρότες, τα κράτη-μέλη, τα... οι ευρωβουλευτές και θέλουν να μάθουν όλοι τι θα κάνω εγώ, τι προτίθεμαι να κάνω για όλα αυτά. Και πρέπει να τα κάνω έτσι ώστε όπως πολύ σωστά είπατε να παραμείνει όλη αυτή η πολιτική ευρωπαϊκή με κοινού στόχους να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό να τηρεί τις αρχές της εσωτερικής αγοράς με ένα κοινό σύνολο στόχων ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτά όλα θα παραμείνουν. Όταν τα κράτη-μέλη ζητούν περισσότερη ευελιξία αυτό σημαίνει ότι πρέπει να του εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις ευελιξίες και όλο το πλαίσιο υλοποίηση και σχεδιασμού μετά το 2020 όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα και τα διάφορα μέτρα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Το συνόλο των κανόνων που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι διπλό μερικέ φορέ. Υπάρχει και σε Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Αντί να έχουμε ένα σύνολο ελέγχων και ένα σύνολο κανόνων, έχουμε δύο. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε κάποια λογική, να σταματήσουμε, να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι του κανονιστικού υπερθεματισμού. Και θέλουμε να προετοιμάσουμε τι σχετικέ ε, προτάσει βάσει των εμπειριών των τελευταίων ετών, ώστε να βρούμε πιο πρακτικού τρόπου υλοποίησης. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη μα και τι νέε τεχνολογίε για του ελέγχους. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπου με τι δορυφορικέ τεχνολογίε που έχουμε και όλε τι τεχνολογίε και τι καινοτομίε που θα έρθουν θα μπορούμε να πραγματοποιούμε πολλούς από τους ελέγχους για αυτές τις συγκεκριμένες πολιτικές και τα προγράμματα με πολύ απλούστερο τρόπο. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική θα συνεχίσει να διαθέτει την ευρωπαϊκή διάσταση της κοινή γεωργικής πολιτικής αλλά η υλοποίηση αυτής της πολιτικής ο επιμερισμός λέει των εργασιών με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλυθεί και να πλουστευτεί προς όφελος των γεωργών και των κρατών μελών. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με το νέο μοντέλο το οποίο θα προσφέρουμε αύριο. Κύριε Σεκέρσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν θέλω να προσθέσω ένα σωρό άλλε ερωτήσει. Ε, θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο ήδη και να υποβάλω και μια ερώτηση. Το πρόβλημα των νέων γεωργών. Ο αριθμός των νέων ε, γεωργών ε, εξαρτάται και από το εισόδημα, από το επίπεδο ε, διαβίωσης, από τη δυσκολία αυτού του επαγγέλματος, από τους κινδύνους που εμπεριέχει, τη δυσκολία πρόσβασης σε αρρώσιμες γέες. Υπάρχουν ένα σωρό ασφάλειες. Ποια θα ήταν η κατάσταση σήμερα αν δεν είχαμε φτιάξει την κοινή πολιτική. Αυτή είναι η μία ερώτηση. θέλω να ξέρω αυτό, σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για τους νέους γεωργούς και πρέπει να παρουσιάσουμε μια πιο μακρόπνοη και οραματική προοπτική στους νέους γεωργούς. Με την παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων για την περίοδο μετά το 2020, σε αυτό το πλαίσιο Ίσως ε, δεν θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για μια πιο μακρόπνοη και διορατική μεταρρύθμιση βλέποντας προς το 2050 σκεφτόμενη την παγκοσμιοποίηση και τις εξωτερικές συνθήκες οι οποίες ε, πάντοτε επηρεάζουν ε, την κοινή πολιτική Αυτό είναι κατανοητό γιατί έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε μια παραγωγή σε χαμηλότερο κλίμακα, έχουμε μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Είναι ένα μοντέλο για το οποίο είμαστε περήφανοι. Όμως τα διεθνή συστήματα είναι πολύ διαφορετικά. Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ανταγωνιστικότητα σε άλλες περιοχές, ε, σε άλλες περιφέρειες, λιγότερη σημασία στην ποιότητα στις περιοχές της Υπέθρου, ας πούμε στον ΠΟΕ ή σε πλαίσιο διμερών συμφωνιών, επικρατούν διαφορετικά στάνταρ. Και οι δραστηριότητες ε, της Κομισιόν είναι σημαντικό να ε, μπορέσουμε να ε, συμβιβαστούμε και να βρούμε λύσει σε διεθνέ επίπεδο. Τώρα, δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η πρόσβαση στις γέες. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις αρρώσιμες γέες. Συχνά οι εκμεταλλεύσεις είναι αντικείμενο κερδοσκοπία. Και... και είναι και μια μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίων. Και αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει εδώ να αντιμετωπιστούν. Και τελευταία ερώτηση Θέλω να μιλήσω για την ασφάλεια, για την απλοποίηση και για την ε, διοικητική διαχείριση. Εγώ είμαι υπέρ της απλοποίησης, όμως ταυτόχρονα πρέπει να σεβαστούμε τα πρότυπα και μια ολόκληρη σειρά κανόνων. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, εντάξει. Αλλά όταν ε, ξεσπάσει μια επιδημία, μια επιζωτία ε, και αρχίσουν να εξαπλώνονται τα μικρόβια και τα βακτήρια, ε, τότε αρχίζουμε να ρωτιόμαστε, μα πού είναι η διοίκηση, με ποιον πρέπει να μιλήσουμε, σε ποιον να απευθυνθούμε. Και ο, και ο φορολογούμενος θέλει να ενημερώνεται πληρώνει. Ε, θέλει να ξέρει ποιε είναι οι υπηρεσίε που του προσφέρουν οι αρχές, πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια παρακολούθηση, μια εποπτεία όλων αυτών των πτυχών. Το 98%, 99% των ε, γεωργών έχουν, πιστεύω, μια προσέγγιση σωστή μέσα στα σύμμορφη με, την, τον νόμο. Ε, υπάρχουν όμως και σπατάλες ή λάθη. Εσείς τι πιστεύετε. Ναι. Κύριε Πίτροπε, ο φορολογούμενος κυρίως θέλει να ξέρει πώς το πρόβλημα των νέων αγροτών λύνεται μόνο με περισσότερα χρήματα. Μας έδειξε το ελεκτικό συνέδριο ότι τα περισσότερα χρήματα αυξάνουν μόνο το εισόδημα. Δεν έχουμε δει ποτέ τέτοιο πρόγραμμα που να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Επειδή ρώτησε ο συνάδελφο, ήθελα να βάλω κι εγώ μια εμβόλυμη ερωτησούλα. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέτε ότι το πρόγραμμα της νέας αγρότης είναι αναποτελεσματικό. Mm. Αυτό επενήσεστε. Ναι, αναμφίβολα οι στηρίξει που δίνουμε στου νέου αγρότε δεν είναι τόσο αποτελεσματικέ όσο θα θέλαμε. Τα νούμερα μιλάνε μόνα του. Μόνο 6% των νέων ανθρώπων κάτω των 40 ε, μπαίνουν στη δραστηριότητα αυτή. Έχετε δίκιο. αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε αυτά τα προγράμματα όσο αποτελεσματικά είναι αποτελεσματικά είναι για να τα κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά διότι υπάρχει μια απέτηση πολιτικής να εμπλακούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι τώρα κατά πόσο αυτό είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωση του κράτους μέλους ε, μείγμα και των δύο θα έλεγα εγώ από φορολογική άποψη είναι πολύ ευκολότερο πιστεύω για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες να προσαρμόσουν τα φορολογικά μέτρα τις φορολογικές ρυθμίσεις ε, ώστε να βοηθήσουν τους νέους να εμπλακούν περισσότερο στις ε, γεωργικές δραστηριότητες. Ε, τα θέματα της πηγής κινητικότητας για παράδειγμα ήταν, έχουν παίξει ρόλο. Μας ανησυχεί το ότι δεν φέρουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Πρέπει να το εξετάσουμε και για τη μεταρρύθμιση μετά το 2020. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κομαγκρή μίλησε για τα ε, πρότυπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Πολύ σημαντικό για τα όσα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εισαγγεί στα μέτρα μας ε, ε, λόγω των τελευταίων ασθενειών που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πολλά μέτρα ιχνηλασιμότητας που δείχνουν στους καταναλωτές και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουμε κάποια κριτήρια και κάποια υψηλά επίπεδα όσον αφορά τα τρόφιμά μας. Επίσης προωθούμε τρόφιμα υψηλής ποιότητας ε, και υπό τη μορφή των γεωγραφικών ενδείξεων ε, και δίνουμε πολλές ε, ευκαιρίες πρόθεσης σε πολλές εταιρείες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηγήσουμε στους καταναλωτές και στην Ευρωπαϊκή σε ολόκληρο τον κόσμο ότι έχουμε φαγητά υψηλής ποιότητας αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο δομέα των φυσικών μας πόρων και της αηφορίας. Η προστασία των φυσικών μας πόρων, ο τρόπος παραγωγής τροφίμων είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάζουμε όλο και περισσότερο σε επόμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ διασφαλίζοντας ότι η γεωργία μας και οι διαδικασίες παραγωγής τροφίμων ε, θα ενοποιηθούν σε όλα αυτά για καλύτερη ε, κάλυψη των διεθνών αναγκών. Και αυτό θα το δούμε αύριο. Τώρα το θέμα της διαχείρισης κρίσεων στο ε, περίπτωση επιβλαβών οργανισμών ή νόσων, πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον. Όλα αυτά θα αποτελέσουν κομμάτι των συζητήσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα ταμείο εντό τη ε, πολιτική ή εκτό πολιτική για όλου αυτού του τομεί που θα επηρεαστούν από κάποια φυσική καταστροφή που θα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, σε πυρκαγιέ, σε πλημμύρε ή από οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κρίσμα, κρούσμα νόσου. Ε, εκεί θα πρέπει να δούμε πού θα ε, διατίθεται κάποιο ταμείο ε, για να εκφραστεί αλληλεγγύη ε, προς τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα απαιτηθεί ενδεχομένως περισσότερη συνεργασία μεταξύ γεωργίας, πολιτικής γεωργικής και πολιτικής περιφερειακής. Η πρόεδρος έχει δίκιο για το όραμα του 2050, αλλά εμείς τώρα μιλάμε για την ΚΑΠΑ από περιβαλλοντική και κοινωνική και οικονομική άποψη παίζει σημαντικό ρόλο και στους τρεις αυτούς τομείς. Ε, οικονομικά τώρα έχουμε μια επιτυχία. Το συζυγείο πληρωμών πολλών κρατών μελών έχει βελτιωθεί σημαντικά όσον αφορά τις εξαγωγές ε, ε, και ειδικότερα στις προγραμματικές χώρες, στη χώρα που γνωρίζω εγώ πολύ καλά, την Πορτοκαλία, για παράδειγμα, την Ελλάδα. Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μνημόνια έχουν δει μεγάλες βελτιώσεις. Περισσότερη απασχόληση, περισσότερες δραστηριότητες το 1 τρίτο των νέων θέσεων εργασίας ε, σε αυτές τις χώρες ε, οφείλεται σε ε, εγγενείς τομείς αγροτικούς. Δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι η γεωργία αποφέρει ωφέλει και οικονομικά. Δεν, είναι, δεν υπάρχει μόνο για κοινωνικούς και για περιβαλλοντικού λόγου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Τώρα, το όρόμα του 2050 σχετίζεται με την αηφορία, τη μετάβαση σε μια βιώσιμη γεωργία. Εκεί θα χρειαστεί να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες ε, για την υλοποίηση των διεθνών συμφωνιών μα. Δυστυχώ θα πρέπει να σας φάω και εγώ λίγο από το χρόνο σας. Ε, θέλω να ανακοινώσω ήδη το εξή. Αύριο στην ανακοίνωσή σα, αν πείτε ότι στο μέλλον όλοι οι έλεγχοι θα γίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους και δεν θα γίνει η Γενική Διεύθυνση. Δεν το κάνει η Γενική Διεύθυνση που κάνει επιτυχώς διορθώσεις. Αυτό θα είναι λόγος για την Επιτροπή μας, όχι ε, ε, να είναι μόνο πάρα πολύ θλιμμένη, αλλά να αναζητήσει επαφή μαζί σας νωρίτερα από του χρόνου τέτοιο καιρό. Οι διορθωτικές εργασίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση βοήθησαν για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές. Δεν μπορεί η γραμμή να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαφίεται στα κράτη-μέλη, το Ελεγκτικό Συνέδριο επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κανεί πια δεν κοιτάει του λογαριασμού. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και θα ήταν πάρα πολύ ε, λυπηρό το νέο αυτό για το φορολογούμε, τον οποίο εμεί εκπροσωπούμε και όχι απλώ ε, θα μας βρείτε αντίθετους, αλλά θα μας βρείτε και σε υποχρέωση να οργανώσουμε την αντίστασή μας σε αυτό. Ε, ερωτήσεις τώρα. Στην ε, έκθεση 16 του 2007, στην ειδική έκθεση μάλλον για την αγροτική ανάπτυξη, είναι μια συστημική και συστηματική έκθεση που ασχολείται ε, με ε, θέματα διαδικαστικά και είναι λίγων σελίδων. Το ΕΖΙ, το Ταμείο, το γενικότερο, το θεωρείται επιτυχία, ασχολείται και με την αγροτική ανάπτυξη υπάρχουν ε, δυσκολίες διοικητικές και προσαρμογής. Αυτό το ταμείο το ευρύτερο είναι επιτυχής υπόθεση ή όχι. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με ε, ε τις πληρωμές. Η Σουηδία έχει 14%, η Γαλλία 10,8%, 11% η Τσεχία, 6,7% η Σλοβακία. Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται προγράμματα δράσης, αλλά συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε προβλήματα. Για ποιο λόγο στις χώρες αυτές. Και μπορείτε να λάβετε θέση συγκεκριμένα. Και μια που κατονομάζουμε χώρες, μας είπατε ότι ο Ουγγρικός Οργανισμός Πιστοποίησης που μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει δήλωση αξιοπιστίας δεν έχει ελέγξει δηλαδή τις πληρωμές του οργανισμού πληρωμών, λέτε ότι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2018 θα το πράξει. Γιατί τέτοια καθυστέρηση. Είναι καλή ιδέα. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την εκτέλεση και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Θα ήθελα να σας εκφράσω την προσωπική μου υποστήριξη για τη σύγκρουση συμφερόντων ε, στην Τσεχία Εκεί ο οργανισμός πληρωμών έχει επικεφαλής έναν ε, ε, βουλευτή, ο οποίος έχει και άλλα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και τα μέτρα για την αγορά είναι πολλαπλά, είναι περίπλοκα, αλλά έχουν και ε, εντυπωσιακά ασφάλματα. 10% στη Γαλλία 9% ε, στα οποροκυπευτικά ε, στον Ίνο και αλλού ε, για μέτρα, τα μέτρα στήριξης αγοράς που έχουν μεγάλα ασφάλματα τι σχέδια έχετε πέρα από τα προγράμματα δράσης πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού υποφέρουμε γιατί όλοι οι έλεγχοι και οι ειδικοί για την πολλαπλή ε, συμμόρφωση τα ρίχνουν στον οικονομικό έλεγχο. Όταν μιλάμε για έλεγχο, δεν είναι πάντα οικονομικός έλεγχος, δεν ισχύει. Πόσο ποσοστό ε, έχουμε λογιστικό έλεγχο και πόσο ποσοστό τεχνικό έλεγχο ε, επί της ουσίας. Επειδή ταξιδεύετε πολύ και τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, στην πολλαπλή συμμόρφωση έχουμε 2,79% κάτω του 3% των δικαιούχων που ελέγχθηκαν επιτόπου. Άρα το 97% δεν ελέγχθηκαν. Γιατί οι διοικητικοί έλεγχοι δεν φτάνουν μέχρι το δικαιούχο. Όταν λέω ότι δεν ελέγχεται τον γεωργικό τομέα, μου λέει ο κύριος Μαγκέλε ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε 100% αλλά θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή ε, στους δικαιούχους και στις κρατικές αρχές ότι το 97% δεν ελέγχεται ε, τους τελικούς δικαιούχους. Αυτοί που ελέγχονται, ελέγχονται δρακόντια και πραγματικά στο κεφάλι, αλλά είναι 3%. Αλλιώς με τέτοιους ελέγχους θα είστε σε αμυντική θέση και θα σας πούνε καταργήστε τελείως τους ελέγχους. Και αν καταργήσουμε τους ελέγχους τότε δεν θα φτάσουμε ποτέ στα αποτελέσματα με βεβαιότητα. Και άλλη ερώτηση. Διάβασα τη συνέντευξή σας το περασμένο Σαββατοκύριακο για το Brexit και την ε, Ιρλανδία. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς αξιολογείτε ε, τις επιπτώσεις στον Ιρλανδικό γεωργικό τομέα ε, του Brexit και τη σχέση με την Βόρεια Ιρλανδία και κατάσταση. Το ξέρω ότι είναι η πατρίδα σας αλλά θα ήταν ενδιαφέρον και για μας να ακούσουμε μερικά πράγματα. Και ένα θέμα το οποίο με απασχολεί εδώ και καιρό και με βασανίζει. Στη Γεωργία έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας που είναι αγρότες ή υπουργοί Γεωργίας παλαιότερα και έχουμε μια μελέτη για τη σύγκρουση συμφερόντων. Η Γενική Διεύθυνση τι κάνει με τους συνομιλητέ σας που είναι σε μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων. Κύριε Σικέρης, και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνονται πράγματα, ε, να ορίζουν ε, ορισμένοι άνθρωποι τους κανόνες και να είναι ταυτόχρονα οι ίδιοι οι άμεση δικαιούχοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς επιτρέπεται. Και τώρα έχετε το λόγο μετά από όλα αυτά που σα ρωτώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας διαβεβαίωσω ότι θα έχουμε πολύ υψηλή εποπτεία και έλεγχο των χρημάτων των φορολογουμένων και όποιος ε, νομίζει κάτι διαφορετικό σφάλει. Τα συστήματα που έχουμε στήσει για να προστατεύεται ο προπολογισμό έχουν αποδείξει και από τη σημερινή συζήτηση ότι αποδίδουν. το σφάλμα είναι χαμηλό, το χαμηλότερο όλων των εποχών και έχουμε εργαστεί προς την αγροτική ανάπτυξη και θα συνεχίσουμε. Εργαζόμαστε πραγματικά πολύ για να μειώσουμε και εκεί το σφάλμα στο δεύτερο πυλώνα. Το μέσο είναι πιο, και το μέτρο πιο στοχευμένο και πιο περίπλοκη η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης και είναι και στη συνυπευθυνότητα και στη χρηματοδότηση. Είναι μεικτή η προσέγγιση, χρειάζεται βελτίωση και το καταλαβαίνουμε όλοι. Η απλούστευση θα βοηθούσε να μειωθεί το σφάλμα, όπως είπα και σε προλαλήσαντα θα προωθήσουμε τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, βοηθάει αυτό και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερικής Ανάπτυξης και όλες ε, τις ε, ενεχόμενες γενικές διευθύνσεις να έχουμε κοινού ε, κανόνες για τη διαχείριση των προγραμμάτων EASY, αλλά τα σημερινά δεν πρόκειται να μειώσουν κάτω της 100 το σφάλμα, κατά την άποψή μου, στο σημερινό πλαίσιο. Χρειάζεται πολιτική να μειωθεί σε λίγους στόχους και λίγα μέτρα για να έχουμε πιο εύκολο έλεγχο. Απ' τη μια θέλουμε περισσότερη δραστηριότητα στην Ήπεθρο με τα προγράμματα και τα μέτρα. Και αν τα μειώσουμε, μάλλον θα έχουμε λιγότερα σφάλματα. Εμείς προσπαθούμε όμως να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία μας ε, για τις επιδόσεις και με χαρά να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Ελεκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή σας ε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους. Για ορισμένες από τις χώρες που αναφέρατε για την Ουγγαρία το 2016 για τη διαχείριση ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί με δήλωση αξιοπιστίας από την αρμόδια αρχή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 20 Φεβρουαρίου αναμένεται με την ετήσια έκθεση για το 2017 και τότε θα εξετάσουμε αυτή την γνωμοδότηση. Δεν έχει έρθει ακόμα. Και μέχρι τότε δεν θα έχουν προταθεί και λογαριασμοί για, για τα οικονομικά για τη Σουηδία και τη Σλοβακία πρέπει να ενημερωθώ περισσότερα. Δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία, θα σα τα στείλω όμω. Ανέφερθηκα προηγουμένω στη Τσεχική Δημοκρατία για τη σύγκρουση συμφερόντων και το ξανασχολιάσατε. Όλα αυτά τα παράπονα και τις καταγγελίες τα σημειώνουμε και τα δρομολογούμε τις διαδικασίες και μεταξύ αυτών και των Όλαφ. Γίνονται έρευνες σε περίπτωση που υπάρχει λόγος και για την τσεχική δημοκρατία δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχο, όπω σα είπα προηγουμένω. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί, θα σα δώσουμε τα στοιχεία. Βεβαίω έχουν ε, ευθύνη και τα κράτη-μέλη για τη σύγκρουση συμφερόντων, για του ανθρώπου που βάζουν υπουργού γεωργία, α πούμε. European level. Ή που συμμετέχουν σε διάφορε συσκέψει σε ευρωπαϊκά φόρα. Τώρα, ένα αγρότη, δηλαδή να μην μπορεί να συμμετέχει ποτέ, να μην είναι μέλος τη Επιτροπής Γεωργίας, τόσο πολύ να το τραβήξουμε το θέμα της σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό νομίζω είναι υπερβολικό, αρκεί να δηλώσει κανείς τα συμφέροντα που έχει ε, βεβαίως ε, να μην έχει κάποια δραστηριότητα παράνομη, απάτε και απιστίες και Και όταν υπάρξει κάποια καταγγελία θα την αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η ισορροπία. Αυτό περιμένουμε να κάνουν οι άνθρωποι για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων. Τα μέτρα για τη στήριξη αγορά και πάλι. Ακούμε ότι υπάρχουν πολλά ασφάλματα. Εκεί και πάλι έμεθα σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Και καταναλώνουμε και, και τα κράτη-μέλη πολλούς πόρους εκεί για να αστυνομεύουν, να παρακολουθούν τους ε, πόρους που δίνουμε. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να επαγρυπνούμε κι εμείς. Μετά με κάνατε μια ερώτηση πάρα πολύ περίπλοκη. Εγώ δεν γνωρίζω τόσα πολλά όσο εσείς για τον οικονομικό έλεγχο και την οικονομική διαχείριση σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση. 5% ελέγχους κάνουμε και άλλους με το ελεκτικό συνέδριο. Και έχουμε ένα σύστημα όπου συνεργαζόμαστε για να δούμε ποιο είναι το υλικό που ελέγχουμε. Μάλλον το, υλικό, το πραγματικό σφάλμα. Και νομίζω καλό πάει σε γενικές γραμμές. Τα συστήματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια αυτό δείχνουν. Όταν βλέπουμε τι γίνεται, ότι οι αγρότες γνωρίζουν τους κανόνες, όπως και τα κρατημέλη γνωρίζουν τους κανόνες. Καμιά φορά δυσανασχετούν, αλλά δεν σημαίνει ότι τους αγνοούν. Και έχουμε συστήματα ελέγχου ε, στη συνδιαχείριση. Θα χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και ε, δορυφορικές για ε, ε, τους τομείς που είχαμε προβλήματα με τα κράτη-μέλη. για να είναι η λύση μόρφωση πιο πιστή προς την πραγματικότητα στο μέλλον. Νομίζω η πολλαπλή συμμόρφωση ήταν ένας μηχανισμός που απέδωσε και σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής το βλέπουμε. Και στο μέλλον θα έχουμε δράσει για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, για την ποιότητα των υδάτων, με απλούστευση, αλλά πάντα τηρώντας τους κανόνες και των χρημάτων που θα παίρνουν οι αγρότες. Δίνουμε χρήματα με όρους. Η αρισιμότητα είναι κάτι που θα αυξηθεί στο μέλλον. Τώρα για το Brexit, να μην σας φάω όλο το χρόνο, θα μπορούσε εδώ συζητάμε, αν αρχίσω δεν να συζητάω και με τον κύριο Φλάνακαν, χαιρετίσματα. Ε, δεν υπάρχουν πάντως ε, καλές ειδήσει ε, από τον Brexit ούτε για την Ελλαδία, ούτε για το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ μεγάλες εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε κοινό χώρο ταξιδίων από το 1991. θα διαταραχθεί πάρα πολύ και η κυκλοφορία και η διοίκηση. Το 48% του συνολικού γεωργικού μας εμπορίου είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στην ίσο της Ιρλανδίας πρακτικά καθημερινά έχουμε 3 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος. Από τη Βόρεια Ιρλανδία καθημερινά ε, καταλήγουν σε γαλακτοκομεία για την επεξεργασία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα έχουμε όταν θα πρέπει να διερχόνται σύνορα μεταξύ Βορρά και Νότου. Είναι σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και είμαστε σε μια δύσκολη ε, εποχή. Περάσαμε από δύσκολη εποχή για να φτάσουμε σε ειρήνη και ηρεμία ε, μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ιλλανδίας αλλά και μεταξύ της νήσου της Ιλλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ε, θέματα επανειλημμένα έχω πει ότι ψήφισαν Brexit οι Βρετανοί για να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι από κάποια πρακτικά μέτρα που ήθελαν να εξακολουθούν να ισχύουν για το εμπόριο και την ελεύθερη διακίνηση ε, μεταξύ των δύο νησιών. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή στην πολιτική διαδικασία και ελπίζω να πριτανεύσει ε, και να συνεχίσει να εκφράζεται η καλή βούληση των υπολείπων 26 προς την Ιρλανδία για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα και το λέω ως Ιρλανδός αυτό. Η κυρία Γκρέσλε, δεν άκουσα την άποψή σας για την ένταξη του ΕΛΑ στο ΕΖΙ, στο ΕΖΙ. We are in discussions at the moment with uh, Commissioner Είμαστε σε διαβουλεύσεις με τις Επιτρόπους Κρέτσου και Τάισεν για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κοινού κανόνες, όχι ενιαίους κοινού ε, στα διάφορα προγράμματά μας και τα μία. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά από πλευρά συνέργειας και συμπληρωματικότητα για να αρθεί κάποια γραφειοκρατία που έχουν τα προγράμματα και στις ε, νομοθετικές προτάσεις που θα φέρουμε το 2018 για την περίοδο μετά το 2020 ελπίζω να δείτε κάποια βελτίωση. The best at the end, και το τελευταίο και καλύτερο τώρα είναι ο κύριος Βόν. Ε, ε, ε, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη, χρειαστήκε να φύγω για να απαντήσω ένα τηλεφώνημα. Οπότε αν επαναλάβω κάποια ερώτηση, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το Brexit. Αυτή την εβδομάδα κάνετε και κάποια σχόλια για τις επιλογές που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα σύνορα με την Ιρλανδία ε, και τις συνέπειες που θα έχουν όλα αυτά για τους Γιώργους ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Συνεχίστε να κάνετε αυτά τα σχόλια διότι πράγματι οι συνέπειες θα είναι σημαντικές και για την Ιρλανδία αλλά και για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε μια προσέγγιση κοινή λογική για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι δύσκολη δουλειά που έχετε. Το να δώσετε στου Γεωργού όσα θέλουν και να εξακολουθούν αυτοί να είναι δυσαρεστημένοι. Είναι πολλά αυτά που έχετε να κάνετε. Είναι δύσκολα. Μια από τι διαμαρτυρίε του σημερινού προγράμματο ε, ήταν το RDP. Πολλά παράπονα, πολλέ διαμαρτυρίε από Γεωργού αλλά και από κυβερνήσει ότι άρχισαν τα RDP πολύ αργά. Ε, και άκουσα πολλά σχόλια λοιπόν. Ε, υπάρχουν κάποια διδάγματα που έχουμε αντιλήσει για το μέλλον. Μετά το 2020 το RDP θα ελπίζω να μην ξεκινήσει τόσο αργά όσο στην προηγούμενη περίπτωση. Το επόμενο ερώτημα για την ευελιξία που δίνουμε στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν ε, τη μεταφορά χρημάτων από έναν πυλώνα σε άλλον. Έχει γίνει ανάλυση καθόλου για όλα αυτά, γιατί ο φόβος εκεί ήταν ότι ορισμένα κράτη-μέλη θα μετέφεραν τόσα πολλά χρήματα από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1 που αυτό θα επηρεάζει τα γενικά αποτελέσματα. Το γενικό καλό, δηλαδή τις βελτιώσεις που θέλαμε να επιφέρουμε στις διάφορες κοινότητες. Έχετε σχόλια γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και το τελευταίο για τους νέους ε, γεωργούς. Πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν. Μιλάμε για μέτρηση των επιδόσεων οι επιδόσει είναι κάτι που μπορούμε να μετρήσουμε. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε είναι ο αριθμό των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται στι γεωργικέ δραστηριότητε. Γιατί όπω ξέρουμε, ε, γεωργοί που έχουν ε, νέα παιδιά και αγόρια και κορίτσια, πολλά παιδιά λένε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν τι γεωργικέ δραστηριότητε ε, μετά τη συνδιεξουδότηση των γονέων του. Αυτό είναι πρόβλημα. Λέτε ότι είναι δύσκολο, πράγματι. Και για το μέλλον τώρα πέραν της επικέντρωσης στους νέους ε, αγρότες ε, σε ηλικία θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στους νέους αγρότες ε, νέους ως δραστηριότητα για τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν γεωργικές δραστηριότητες χωρίς να τις κληρονομούν να δούμε πώς αυτό διαμορφώνει το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση uh, Ευχαριστώ κύριε Βον ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις Ξέρω ότι το θέμα σας αφορά ιδιαίτερα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ε, από τη φύση τους ε, ξεκίνησαν αργά διότι λόγω της χρηματοδότηση των προγραμμάτων ε, καθυστέρησαν δημοσιονομικά και λόγω των κρατών μελών και των περιφερειών. Είναι πραγματικότητα. Το 23-24% είναι η απορρόφηση των ταμείων αυτών αυτή τη στιγμή και επιταχύνεται μάλιστα όσον αφορά την υλοποίηση. Έχουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο έτος, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να πάνε σε τομείς που δεν να, όπου δεν προτίθεται να πάνε στην αρχή του προγράμματος. Αναγνωρίζω ωστόσο τα όσα λέτε ε, όσον αφορά τα νούμερα, αλλά αυτή είναι η φυσιολογική τροχιά Και όπως είδαμε και από τα τελικά αποτελέσματα από το περασμένη προγραμματική περίοδο είχαμε και φτάσει σε 96-97% απορρόφησης. Οπότε αυτό που μου λένε ότι 22,6% είναι ε, το FRD. Ε ε, ξέρω ότι κάποια άλλα προγράμματα ακόμα είναι σε μονοψήφια ποσοστά, αλλά λαμβάνουμε υπόψη τα όσα λέτε. Τώρα τη μετακίνηση των χρημάτων από τον πυλώνα 2 στον 1 μια-δυο χώρες ε, το παρατράβηξαν λίγο από ό,τι ξέρω. Πρέπει να το εξετάσουμε βλέποντας ποιοι είναι οι στόχοι, του, για μετά το 2020. Θα λαμβάνουμε πέρα των στόχων υπόψη και τις επιδόσεις τώρα. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τέτοιες μετακινήσεις χρημάτων από τον πλώνα 2 στον πλώνα 1 γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά καλά πράγματα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης ε, και ειδικότερα στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα και τις υπηρεσίες. Και πολλοί νέοι αγρότες ασχολούνται με αυτά. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν προγράμματα ώστε να συμβούν όλα αυτά. Αλλιώς ε, όμως αν αφαιρέσουμε χρήματα από τον πλέον 2 δεν θα φέρουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Με ενδιαφέρον αυτό που είπατε όχι μόνο για τους νέους σε ηλικία αγρότες αλλά και για τους ε, νέους αγρότες ως ανθρώπους που έρχονται στο επάγγελμα. Αυτό το ηλικιακό όριο είναι λίγο αυθαίρετο. Μπορεί να θεωρήσουν κάποιοι. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον όταν μπαίνουν ε, άνθρωποι ε, στη δραστηριότητα αυτή, ε, πιο μορφωμένοι παλιότερα όταν ήταν κάποιος ε, γιο ε, Γεωργού δεν είχε και πολλέ επιλογέ για να βγει από αυτό αλλά σήμερα ο κόσμο έχει επιλογέ. αλλά υπάρχει μια ομάδα νέων ανθρώπων ε, από οικογένειε γεωργών που ενδεχομένω θέλουν να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση στον αγροδιατροφικό τομέα διατηρώντα λοιπόν τη σχέση με τη γεωργία αλλά όχι όντα καθημερινά γεωργή. Το βλέπουμε και αυτό και στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες ως νέοι άνθρωποι που είναι παιδιά γεωργών και που θέλουν να παραμείνουν στη γεωργία μέσω του αγροδιατροφικού τομέα και σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αντί για γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο τέλος. Ο κύριος Μιλιώνης θέλει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να πω τελειώνοντας ότι συμφωνούμε με τον ε, εισηγητή κύριο Σέλερ ότι χρειάζεται καλύτερη προ, ε, προώθηση όσον αφορά την κατανομή των, των κονδυλίων. Σημειώνουμε τα σχόλιά του για τις εξαγωγικές αγορές. Συντόμως ε, θα ξεκινήσουμε έλεγχο για την τα μέτρα μάλλον σταθεροποίησης των εισοδημάτων. Εκτιμώ τα σχόλια πολλών ευρωβουλευτών όσον αφορά τα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου συμφωνούμε ότι πρόκειται για τομέα κλειδί για τη μελλοντική μας εργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο Φλάναγκαν. Κομμουνιστής δεν είμαι. Ε, πολύ περισσότερο που έχω ζήσει σε μια χώρα που είχε ως κρατικό στόχο τον κομμουνισμό. Και στη Γεωργία, το ξέρω, το είδα από τον πεθερό μου τον ίδιο, που ήταν αγρότης από παράδοση αλλά και από μεράκι. Και στην αρχή της δεκαετίας του 60 απαλωτρίωσαν και τις γέες του και τα ζώα του και τα δώσανε σε κρατικές εταιρείε και εκμεταλλεύσεις. Και η Γεωργία ε, στην στην Ανατολική Γερμανία, είχε προσανατολισμό ε, βιομηχανική γεωργία κατά το σοβιετικό πρότυπο με τεράστιες ε, εκτάσεις ανεξαρτήτως οικολογικών καταστάσεων τις καλλιεργούσαν εκεί. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ήταν όμοιρος στη ε, χημική βιομηχανία ήταν αναγκασμένες να αγοράζουν τα προϊόντα τα χημικά και να τα ρίχνουν στα χωράφια που δεν είχε μεγάλη σχέση ούτε με βιωσιμότητα, ούτε με βελτίωση, ούτε με διαφύλωση του περιβάλλοντος. Και τώρα ας κάνουμε τη γέφυρα προς τη σημερινή κατάσταση όπου συμβαίνουν αντίστοιχα βέβαια με προϋποθέσεις οικονομίας της αγοράς. Και θα πρέπει από την Ανατολική Γερμανία να τα πω αυτά, αλλά όχι μόνο ως Ανατολικό Γερμανός. Γεωργικές εκτάσεις και γεωργικά προϊόντα, θα είπε και ο συνάδελφος ε, Σικέσκι, και το τόνισε, είναι αντικείμενο πλέον σπέκουλας, κερδοσκοπίας. Οπότε όταν συζητάμε εδώ για νέους αγρότες ή για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα, το οποίο επάγγελμα ε, προποθέτει και κάποιες συμπεριφορές και κάποιο μεράκι. Το κάνεις και από, από δεν το κάνεις μόνο από επάγγελμα. Ε, έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τώρα των γεών τα τελευταία χρόνια. Με μαζική παραγωγή να είναι ο κανόνας για να ε, περιορίζονται και συμπιέζονται οι τιμές. Οπότε πώς να εγκατασταθεί ένας νέος αγρότης εκεί, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η ζωή του. Παρόλα αυτά, και μάλιστα ε, ε, στην Ανατολική Γερμανία τώρα στα νέα κρατήδια έχουμε δύο γεωργικές ενώσεις από τη μια εκεί που είναι παραδοσιακοί ε, αγρότες, οικολογικοί, με αηφορία και βιωσιμότητα και τους άλλους, τους πιο βιομηχανικούς. Αυτό θα είναι πρόκληση και για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζητήση για τον προπολογισμό επέβαλε το 2018 να υπάρξει αύξηση των πόρων περαιτέρω για τους νέους αγρότες. Αλλά το χρήμα δεν είναι το παν σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και το περιβάλλον έτσι ώστε ε, το επάγγελμα του αγρότη να είναι κάτι ελκυστικό για νέους και λιγότερο νέους. Η συζήτηση έχει ανοίξει, συνεχίζεται και ε, πιστεύω ότι και εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε η Πρόεδρος, να δούμε τι γίνεται με τα μέσα για την αγροτική ανάπτυξη και να τα ε, συνδέσουμε με τα, τους άλλους πόρους το Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης, το EASY, γενικότερα να συνδυαστούν γιατί έτσι θα έχουμε μια εδαφική προσέγγιση και όχι κατακαιρματισμένη και χωριστή. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Μιλιώνη και τους συναδέλφου του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο Χόγκαν και τους συνεργάτες του για τη συζήτηση, για τα στοιχεία που μας έδωσαν για το έργο τους και βεβαίως σας ευχαριστώ και πάλι τους συμβούλους της γραμματείας της πολιτικής μου ομάδας και το βοηθό μου, τον Λούκας Ράιχε. Χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών δεν θα μπορούσα να είχα κάνει ε, τη δουλειά αυτή ως Σας Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε. Επίτροπε που ήρθατε, να ανταλλάξουμε απόψεις, παραμείνατε και περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, γιατί βλέπετε ότι σας έχουμε ανάγκη εδώ ε, να συζητάμε. Εξαρτάται από αύριο, από αυτό που θα πείτε, δεν σας υπόσχομαι ότι θα τα ξαπούμε του χρόνου, μπορεί και νωρίτερα. Σημείο 9. Μελέτη με θέμα μεταβατικές αποζημιώσεις για πρώην αξιωματούχο Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπερβολικά λίγε προποθέσει. Ε, κα, καλωσορίζω την εταιρεία ε, που έκανε τη μελέτη. Και τώρα παρακαλώ μην κάνετε τόσο σάλο εδώ. Ε, παρακαλώ να αποχωρήσετε ε, και αθορύβος. Το λόγο ε, έχουν οι συντάκτες της μελέτης για να την παρουσιάσουν. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλε που μας καλέσατε σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Δεν είμαι βέβαιος κύριε μα θέλετε εσείς να ξεκινήσετε ή εγώ. Εγώ, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας καλέσατε σε αυτή τη μελέτη που αφορά τις μεταβατικές ε, επιδόματα ε, για τους πριν αξιωματούχους και θα αρχίσω να φωνάζω για να μ' ακούτε από κοινού με τον συνάδελφο Κρίστοφ Τέμκε θα προσπαθήσω σύντομα να σας δώσω μια γενική εικόνα του τι είναι αυτές οι μεταβατικές αποζημιώσεις και θα αναφερθούμε σε κάποια θέματα κλειδιά όπως ας πούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι μεταβατικές αποζημιώσεις, ποιος τις παίρνει, για πόσο καιρό, ε, ποιος είναι ο προπολογισμό που ε, χορηγείται και τι συμβαίνει στη διάρκεια το περίοδου ε, του δικαιώματος Αυτό Πρόκειται για μια ε, γενική ε, εξέταση το τι ακριβώς είναι οι μεταβατικές αποζημιώσεις. Μετά θα σας μιλήσουμε για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα διάφορα κράτη-μέλη, στις τρίτες χώρες, στις ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, που επίσης ε, προβλέπουν ε, μεταβατικές αποζημιώσεις. Η ιδέα είναι να επιστήσουμε την προσοχή σας εάν ποτέ θεωρήσετε την ενδιαφέρουσα η μεταρρύθμιση ε, κάποιων πτυχών του συστήματος που ισχύει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αυτή η μελέτη να αποτελέσει ενδεχομένως πηγή έμπνευσης. Now, um, first point of the um, overview, what are transitional allowances? Um, um... Λοιπόν, όσον αφορά τις μεταβατικές αποζημιώσεις, ξέρετε ίσως ότι πρόκειται για πληρωμές που καταβάλλονται σε πρώην μέλη των διαφόρων θεσμών για μια κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τώρα αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με το μάκρος της υπηρεσίας, με τη διάρκεια της υπηρεσίας και όλα αυτά περιγράφονται μέσω, σε ένα ε, αρκετά περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχουν ε, τα διάφορα θεσμικά όργανα και ακολουθούν ε, διάφορες διαδικασίες. Εδώ έχουμε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την απόφαση 2005 2005-684 εδώ προβλέπεται τα συνταξιδοτικά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τους άλλους οργανισμούς υπήρξε μια μεταρρύθμιση το 2016, όπου εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές και άρα τα μέλη του Συμβουλίου της Επιτροπής του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, του Ombudsman, του, ο, ο ας πούμε, Ευρωπαίος υπόπτης για τα δεδομένα, Έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με το αν τα μέλη τοποθετήθηκαν πριν ή μετά το Μάρτιο του 2016 που έγινε και η τελευταία αυτή μεταρρύθμιση. εν συντομία εξετάσαμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Uh, um, um, και εδώ υπάρχουν επίσης ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία είναι βασισμένα ε, στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τα άλλα θεσμικά όργανα. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θέσαμε είναι γιατί υπάρχουν μεταβατικές αποζημιώσεις και περί τίνος πρόκειται. Ε, στόχο έχουν να καλύψουν κάποια οικονομική ανασφάλεια που μπορεί να ζήσουν κάποιοι αξιωματούχοι όταν φτάσει στο τέλος η θητεία τους το ισχύον ε, ρυθμιστικό πλαίσιο το καλύπτει αυτό γιατί η οικονομική ανασφάλεια αναφέρεται ως το, η λογική ε, που διέπει αυτές τις ρυθμίσεις ή όπως κάποιες συζητήσεις που είχαμε με εκπροσώπους των θεσμών ε, έδειξαν ότι πρόκειται και για μια σχέση με στόχο την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων ώστε δηλαδή πρώην μέλη, ε, πρώην αξιωματούχοι πριν ε, φτάσει το τέλος της θητείας τους να αναζητούν επασχόληση σε τομείς ε, όπου μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι μια μεταβατική αποζημίωση θα τους βοηθήσει να μην το κάνουν αυτό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ιστορικό των μεταβατικών αποζημιώσεων, το, τα αρχαία του Συμβουλίου ήταν εξαιρετικά οήθημα, μας καθοδήγησαν στην πρώτη σύνταξη των μεταβατικών αποζημιώσεων. Έχουμε την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων το 1951, όταν ε, για τα μέλη της ε, ΕΚΑΧ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνδρακα και Χάλιβα, δημιουργήθηκαν τέτοιες αποζημιώσεις και χορηγήθηκαν για μια τριετή περίοδο. Ο συνάδελφος Κρίστοφ θα μπει στο βάθος αυτών των θεμάτων, δηλαδή ποια είναι η ιστορία και τεκμηρίωση για αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή οικονομική ασφάλεια και σύγκρουση συμφερόντων και μετά θα συνεχίσω και εγώ. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Πριν πάμε σε αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το ζήτημα. Ουσιαστικά μιλάμε για περιορισμούς μετά την απασχόληση από το 1951. Και μιλάμε ότι υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μεταβατικές αποζημιώσεις από το 1961. Δηλαδή σχεδόν 70 χρόνια το ένα και σχεδόν 55 το άλλο. Το λέω αυτό διότι ως ερευνητής κατά τη διεξαγωγή της μελέτης το βρήκα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι άνθρωποι σαν εμάς ε, πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί που ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα, διοικητικά ζητήματα, γνωρίζουμε πολλά για τους πολιτικούς, μας συναρπάζουν οι αξιωματούχοι, οι σταδιοδρομίες τους, τα σκάνδαλα, οι κρίσεις, τα πολιτικά συστήματα, η λήψη αποφάσεων, ε, τα θεσμικά όργανα. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αλλά δεν γνωρίζουμε καθόλου τι γίνεται μετά, αφού φύγουν από την πολιτική ζωή οι πολιτικοί. Δεν έχουμε στοιχεία καθόλου για το τι κάνουν οι αξιωματούχοι, οι πολιτικοί αφού αποσυρθούν από την πολιτική. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κι άλλο ένα φαινόμενο. Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τις μεταβατικές αποζημιώσεις. Δεν έχουμε βρει ούτε μία μελέτη, ούτε μία συγκριτική μελέτη για τις μεταβατικές αποζημιώσεις. Δεν υπάρχει έρευνα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Δεν έχει γίνει έρευνα όσον αφορά τη χρήση της μεταβατικής αποζημίωσης και δεν έχει γίνει καθόλου έρευνα για τις ανάγκες ύπαρξης μεταβατικών αποζημιώσεων. Στην ακαδημαϊκή έρευνα Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένα σημείο συμφωνίας ότι οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι αιτιολογούνται, ότι είναι εύλογες, ε, νομιμοποιούνται διότι οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης και πρέπει να αποζημιώνονται για τη σκληρή τους δουλειά. Ειδικότερα λόγω του ότι δεν υπάρχουν επιδόματα ενεργείας για πολιτικούς. Λόγω αυτού λοιπόν νομιμοποιείται η ύπαρξη μεταβατικών αποζημιώσεων. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα. Ο είναι ότι η λογική των κανονισμών του 2016 και του 2022 του 67 είναι ότι νομιμοποιείται όλο αυτό ω αποζημίωση για οικονομική ανασφάλεια. Διαβάζοντα λοιπόν αυτά τα έγγραφα μαθαίνουμε ότι οι μεταβατικές αποζημιώσεις ε, για τους πολιτικούς μετά από την αναχώρησή τους θα πρέπει να καταβάλλονται ώστε να αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι για ε, εποχές οικονομικής ανασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες έρευνες για αυτό το ζήτημα, όχι πολλές όπως είπα, αλλά αυτές που υπάρχουν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που να υποστηρίζει τέτοιου είδους αξίωση και τέτοιου είδους ισχυρισμό. Ελάχιστοι πολιτικοί βιώνουν ε, ανασφάλεια, οικονομική φτώχεια. Οπότε αυτό πιστεύουμε είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Νομιμοποιούνται μένει τα μεταβατικές αποζημιώσεις, φυσικά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η βασί της λογικής του ρυθμιστικού πλαισίου οι μεταβατικές αποζημιώσεις απαιτούνται για την αποζημίωση των αποχωρών των πολιτικών σε εποχές ε, οικονομικής ανασφάλειας οι οποίες όπως δεν υπάρχουν. Αυτό πιστεύω στο εγγύς μέλλον θα αναδείξει ένα πολύ βέστο πρόβλημα Πολύ απλό. Το όλο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως το βλέπουμε εμείς, δεν βασίζεται σε αυτά στοιχεία, σε γεγονότα. Δεν νομιμοποιείται, για να σας το πω και έτσι. Και μετά έχουμε επιπλέον ισχυρισμούς, επιπλέον κανόνες σε αυτό το πλαίσιο. Για παράδειγμα, να επιτρέπεται σε επίσημου δικαιούχου, σε αξιωματούχου, σε πολιτικού, αφού αναχωρήσουν, αφού αποχωρήσουν, να του δώσουμε το δικαίωμα να ετηθούν ε, αποζημιώσει παρότι έχουν βρει ήδη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, διότι πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα το κοινό και τα μέσα που επιδεικνύουν ιδιαίτερη αυστηρότητα προς πολιτικούς θα στραφούν προς αυτά τα ζητήματα και θα αρχίσουν να επικρίνουν αυτή την εικόνα του πολιτικού που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Απαιτείται λοιπόν επίγουσα αναθεώρηση του πλαισίου αυτού και τον, να βασίζεται αυτό το πλαίσιο σε στοιχεία, σε γεγονότα. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κριστόφ. Για να συνεχίσουμε την επισκόπηση, το επόμενο σημείο είναι ποιο ουσιαστικά δικαιούται μεταβατικές αποζημιώσεις. Σε αυτό το διαγραμμα πίτας βλέπετε τα ποσοστά στα διαφορετικά όργανα. Φυσικά το μεγαλύτερο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των 750 μελών του, αλλά και οι δικαστή εισαγγελείς ε, όλοι αυτοί στο δικαστήριο επίσης ε, ε, δικαιούνται ε, τα 28 επίτροποι, τα 28 μέλη του ελεκτικού συνεδρίου και η αξιωματούχοι κάποιων άλλων θεσμικών οργάνων ο Ευρωπαίος Υπόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής αλλά και τα 15 μέλη των εκτελεστικών δομών της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για πόσο καιρό διατηρούν το δικαίωμα αυτό οι δικαιούχοι, όπως είπα έγινε μια μεταρρύθμιση σημαντική το 2016 με μια μεγάλη αλλαγή η οποία συνίστατο στη μείωση της μέγιστης διάρκειας των μεταβατικών αποζημιώσεων. Αυτό που βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα είναι με μαύρο χρώμα την μέγιστη διάρκεια των μεταβατικών αποζημιώσεων στα διάφορα θεσμικά όργανα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση. Με κόκκινο χρώμα βλέπετε τη διάρκεια των περιορισμών απασχόλησης για τα διάφορα όργανα. Δύο μηνύματα πρέπει να μας μείνουν από αυτό το διάγραμμα. Πρώτον, το ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές, όπως είπα, έγινε μείωση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ε, όσον αφορά τη διάρκεια των μεταβατικών αποζημιώσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να είναι 36 μήνες, σε άλλα θεσμικά όργανα έχει μειωθεί σε 24 μήνες. Και το άλλο ενδιαφέρον μήνυμα που διακρίνουμε εδώ είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της διάρκειας των μεταβατικών αποζημιώσεων και των περιορισμών απασχόλησης ε, μετά από την αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε ορισμένα θεσμικά όργανα λοιπόν έχουμε το σενάριο που η διάρκεια των μεταβατικών αποζημιώσεων είναι πολύ μεγαλύτερη. Για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον Πρόεδρο της Κομισιόν και για άλλα θεσμικά όργανα φαίνεται τα πράγματα να είναι αντίστροφα. Δηλαδή μετά το 2016 θα έχουμε το Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που θα έχουν 36 μήνες ε, μεταβατικών αποζημιώσεων, ε, συγγνώμη, ε, περιορισμών απασχόλησης αλλά μόνο οι 24 μήνες θα είναι η μέγιστη διάρκεια των μεταβατικών αποζημιώσεων. Τι τιμή έχουν όλα αυτά. Η έκθεση δίνει ένα παράδειγμα ενός αξιωματούχου που έχει υπηρετήσει για πέντε χρόνια στο θεσμικό του όργανο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός μεταφράζεται σε 50.000 ευρώ επί εξαμήνου μεταβατική αποζημίωση σε άλλα θεσμικά όργανα κυμαίνεται από τα 20 μέχρι 30.000 ευρώ ε, σε διάστημα δύο ετών. Πώς μεταφράζεται αυτό σε δαπάνη προϋπολογισμού. Σε αυτό το διαγράμμα βλέπετε με μπλε χρώμα το, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με κόκκινο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις σχετικές δαπάνες. Και οι μαύρες κάθετες γραμμές είναι ε, τα έτη των ευρωεκλογών ε, και ανανέωση της Κομισιόν όπως ε, αναμένεται εκεί πάντα έχουμε από το μια αύξηση ε, του προϋπολογισμού τα χρόνια αμέσω μετά τις εκλογές. Καταλήγοντας το ποσό λίγο πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ μετά από τις τελευταίες ευρωεκλογέ. Τελευταίο σημείο για την επισκόπηση. Τι γίνεται κατά τη διάρκεια του δικαιώματο, υπάρχει κάποιο καθήκον ενημέρωσης. Πρέπει δηλαδή το πρώην μέλος να είναι σε επαφή με το θεσμικό του όργανο και να αναφέρει ποια είναι η κατάσταση απασχόλησής του. Γιατί, διότι ε, αυτή μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό των μεταβατικών αποζημιώσεων. Το υποθετικό σενάριο λοιπόν ως πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε περίπτωση που κάποιο απασχοληθεί σε κάποιο άλλο θεσμικό όργανο ή σε κάποιο άλλο δημοσιο αξίωμα, ο γενικός κανόνας προβλέπει αντιστάθμιση, μείωση ουσιαστικά, ενώ δεν επηρεάζεται η σε καποιο αλλο δημοσιοαξιωμα ο γενικος κανονας προβλεπει αποζημίωση αν απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα το πρώην μέλος για τα άλλα θεσμικά όργανα, οι μεταβατικές αποζημιώσεις τερματίζονται σε περίπτωση απασχόλησης σε άλλο θεσμικό όργανο και αντισταθμίζονται σε περίπτωση απασχόλησης σε οποιαδήποτε άλλη επικερδή δραστηριότητα όπως αναφέρεται στον κανονισμό, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτική. Το επόμενο τώρα, η έκθεση προσπαθεί να δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την προσέγγιση ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών όπως η Ελβετία και ο Καναδάς σε διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ε, δηλαδή ε, και, και διάφοροι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί πώς χειρίζονται ε, τι μεταβατική, τις για να βρούμε κάποιες ιδέες να σας δώσω κάποια παραδείγματα στην Ισπανία και στον Καναδά για παράδειγμα υπάρχει ρητά σχέση μεταξύ μεταβατικών αποζημιώσεων και περιορισμών απασχόλησης σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακαλύψαμε ότι η διευθέτηση όπου ένας πρώην αξιωματούχος παρετείται εθελούσια τότε οι μεταβατικές αποζημιώσεις τερματίζονται αυτόματα. Γίνεται δηλαδή διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορών τρόπων αποχώρησης. Στη Σουηδία και στην Ελβετία έχουμε ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο στην κάθε χώρα όπου οι μεταβατικές αποζημιώσεις ε, ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες ε, των πρώην αξιωματούχων ε, στη Σουηδία και με την ηλικία του. Σε άλλες χώρες δεν απαιτείται ιδιαίτερη παρακολούθηση διότι γίνεται μια εφάπαξ καταβολή στο τέλος της υπηρεσίας. Αυτό συμβαίνει στον Καναδά, στην Τσεχική Δημοκρατία, στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία. Στις κάτω χώρες έχουμε ένα μοντέλο που παρέχει κίνητρα σε πρώην αξιωματούχους να αναζητήσουν ε, νέα απασχόληση. Και μετά σε πολλές χώρες ε, οι μεταβατικές αποζημιώσεις τερματίζονται αυτόματα ανεξάρτητα από τη νέα απασχόληση του πρώην αξιωματούχου. Και τέλος υπάρχει ένας ενδιαφέρον μηχανισμός ε, στην Ισπανία Γι' αυτό το θέμα της αναφοράς ε, ε, οποιονδήποτε αλλαγών στην κατάσταση απασχόλησης και για να αποφεύγονται ασφάλματα, ουσιαστικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενημερώνει την αρμόδια διοίκηση για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση απασχόλησης του πρώην εξωματούχου. Ξαναδίνω τον λόγο στον Κριστόφ. Ευχαριστώ Ρολάντ. Ε, στις συστάσεις θα είμαι σύντομος. Δεν έχουμε αρκετό χώρο για να τις συζητήσουμε όλε. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ε, πολύ κατακαιρματισμένο. Ε, είναι πολύ δύσκολο να το ε, αιτιολογήσουμε όλο αυτό. Τα δικαιώματα διαφέρουν και αυτό είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί, αλλά και η διάρκεια διαφέρει και αυτό δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε. Εκεί υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε να αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ. Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο τα δικαιώματα μπορούν να μειωθούν αν κάποιο απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχίζονται. Και θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να αιτιολογηθεί όλο αυτό. Θα πρότεινα λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε το πλαίσιο. Αυτό που είπα προηγουμένω που για μας είναι το σημαντικότερο. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο βασισμένο σε γεγονότα σε αυτά στοιχεία. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι περισσότερα ε, στοιχεία για το όλο ζήτημα, περισσότερη έρευνα. Για παράδειγμα, κατά βάση δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους λόγους και πώς σχετίζονται οι μεταβατικές αποζημιώσεις με τις συγκρούσεις συμφερόντων πώς αυξάνονται, μειώνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα αυτά είναι καθαρά... Ε, όλα τα σενάρια που μπορούμε να φανταστούμε είναι υποθετικά και αυτό δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο σε αυτό, στις κανονιστικές ρυθμίσεις. Επίσης, ε, πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να εξετάσουμε καινοτόμε μεθόδους και ιδέες. Όπως έχουμε δει σε ορισμένες χώρες, ε, χρησιμοποιούνται μεταβατικέ μεταβατικές ω ως κίνητρα για εξέβρεση νέα απασχόληση. Γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί να μην καταβάλουμε τι αποζημιώσει μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη, αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί να μην τι ε, μειώνουμε μετά από ένα διάστημα, ώστε να παρέχουμε κίνητρα στον πρώην να βρει νέα απασχόληση. γιατί να μην κάνουμε κάτι που έχουμε δει πολλές φορές οι υψηλά ιστάμενους πολιτικούς όταν ε, αντιμετωπίσουν δύσκολες εποχές αφού φύγουν από τη θέση τους γιατί να μην αντικαταστήσουμε τα οικονομικά κίνητρα με άλλα κίνητρα όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπαίδευση. Έχουμε ε, και στοιχεία που μας λένε ότι η ζωή, η συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη ε, όταν αποχωρήσουν. Εδώ έχουμε εστιαστεί μόνο στα οικονομικά κίνητρα, αλλά όχι στα άλλα κίνητρα. Επίσης προτείνουμε να σκεφτούμε το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει να καταβάλλεται ε, προσωρινή αποζημίωση σε περίπτωση θελούσες αποχώρησης. Οι περισσότεροι κανόνες ε, προβλέπουν ότι καταβάλλεται τέτοια αποζημίωση σε περίπτωση εθελουσίας αποχώρησης και αυτό ε, για ορισμένους αποτελεί πρόβλημα. Τέλος, και δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε τώρα, θεωρούμε ότι αν πάμε πίσω στο 1951 όπου οι περιορισμοί απασχόλησης μετά από τη θητεία υπήρχαν, σήμερα πλέον έχει έρθει η ώρα να ευθυγραμμίσουμε τους περιορισμούς αυτούς και με τις περιόδους καταβολής των μεταβατικών αποζημιώσεων. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ αυτών των δύο. Και φυσικά και η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της παρακολούθησης των πληρωμών αυτών. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο μας υποβλήθηκε όταν συζητήσαμε με τους διάφορους θεσμούς, ότι δηλαδή ήταν δύσκολο να κρατάμε επαφή με τους πρώην αξιωματούχους, ότι, υπάρχει, ότι βασικά υποφιόμεθα στην καλή πίστη όσον αφορά τις αιτήσει δηλώσεις και εν γέννη τα πράγματα λειτουργούν καλά, όμως έχουν υπάρξει ε, σφάλματα και... Ε, προβλήματα και γι' αυτό θα πρέπει να ζητηθεί να συμπληρώνεται μία ετήσια η δήλωση στην εφορία για να μπορούμε εμείς να επαληθεύσουμε και να αποφύγουμε οποιοδήποτε σφάλμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, με τόση χαρά μας δώσετε για τόσα λίγα λεφτά. Μπράβο, ευχαριστώ. Ε, αναφερθήκατε ε, σε αξιωματούχους και βάλατε στο ίδιο τσουβάλι κατόχους εντολής και κατόχους και θητείας. Δηλαδή, υπάρχουν, στη Γερμανία γίνεται πολύ σαφή διάκριση ανάμεσα στους βουλευτέ, αυτούς που έχουν μια εντολή και σε κάποιου αξιωματούχου που έχουν θητεία. Και μάλιστα μέχρι και ποινικό σημείο πούμε, γίνεται η διάκριση αυτή. Εσεί γιατί τα ανακατέψατε αυτά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να μην ε, προκαλέσουμε σύγχυση και πραγματικά μιλούμε για διαφορετικές ε, νομοθετικές ρυθμίσεις για διάφορους ε, τομείς Τώρα στην παρουσίαση που μιλάμε για αξιωματούχους μπορεί να προέκυψε κάποια σύγχυση, αλλά έχετε δίκιο. Η έκθεση επιμένει στη διαφορά ότι άλλο είναι να έχεις μια εντολή, να είσαι δηλαδή ευρωβουλευτής και άλλο να είσαι αξιωματούχος ε, διορισμένος για κάποιο διάστημα, για κάποια θητεία ε, σε ένα θεσμικό όργανο. Το βλέπουμε και από τη βιβλιογραφία αυτό, γίνεται σαφής διάκριση. Um, ε, δεν ε, το συγχαίουμε καθόλου. Και μας ζήτησαν να κοιτάξουμε και, τα δύο, και τις δύο κατηγορίες, και πρώην ευρωβουλευτές αλλά και πρώην αξιωματούχους διορισμένους. Μάλιστα. Ο κύριος ε, εισηγητής, ο κύριος Σάβαρμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ ειλικρινά στο τμήμα μελετών του Κοινοβουλίου και τους ερευνητές, τον κύριο Μπλόμαγερ και τον κύριο Ντέμκε, που μας ε, έδωσαν αυτή την επισκόπηση, πολύ ενδιαφέρουσα, για ένα θέμα που το θεωρώ μάλλον σημαντικό. Πραγματικά έχει έρθει η ώρα, πιστεύω, να εξετάσουμε σε βάθος αυτό το εκρεμές ζήτημα που αφορά την δημοκρατική διακυβέρνηση και τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προπολογισμού της. Και δεν είναι μόνο αυτό, πολύ περισσότερο είναι το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εικόνα που δίνουμε στα μάτια του πληθυσμού. Μελέτησα τις διατάξει που ισχύουν για τι μεταβατικέ αποζημιώσεις πρώην Ευρωβουλευτών, μελών τη Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων υψηλών βαθμών αξιωματούχων. Πάρα πολύ σημαντικό. Είδα ότι πρόσφατα είχαμε ανησυχητικά παραδείγματα όπου πρώην αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε καθήκοντα σε άλλη δημόσια υπηρεσία, εξακολουθώντα να λαμβάνει σημαντικά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή μεταβατικών αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η νομική βάση και η διακυβέρνηση αυτών των αποζημιώσεων θα πρέπει να είναι άψογη, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την νομιμοποίησή τους. Δείχνει η μελέτη ότι τέτοιου είδους αποζημιώσεις είναι μεν κοινέ αλλά και νομιμοποιούνται και εύκολα. Αλλά ταυτόχρονα εμπίπτουν σε κάποιες διατάξεις και όρους κάπως ρηχούς. Τι εννοώ, ότι επαφείται στην καλή βούληση και στην ευθύνη του ίδιου του δικαιούχου να εξασφαλίσει ή να διασφαλίσει ότι ακολουθεί τους κανόνες και δείχνει την απαραίτητη συμμόρφωση. Όπως μάθαμε, οι ε, μεταβατικές αποζημιώσεις δεν είναι ε, κάτι το οποίο στερείται ατασταλιών και σφαλμάτων. Σημειώνω τις συστάσεις της μελέτης, συμφωνώ. Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και αναθεώρησης με βάση ε, τα στοιχεία, όπως είπε ο κύριος Ντέμκε. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες για όλους τους αξιωματικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν μεταβατικές αποζημιώσεις και βεβαίως να εξακριβώνουμε και να ελέγχουμε ότι πληρώνονται, καταβάλλονται αυτές οι αποζημιώσεις μόνο όταν χρειάζεται και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι τώρα αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε με βάση αυτή τη μελέτη, η οποία είναι πολύ καλή, και με εκπλήσει πάρα πολύ αυτό που άκουσα ότι είναι η πρώτη ακαδημαϊκή δουλειά που γίνεται έτσι, όλων των εποχών. Απίστευτο. Τώρα όμως που έχει μελετηθεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να το λάβουμε ως βάση τη συγκεκριμένη μελέτη και να διαρευνήσουμε περαιτέρω το φαινόμενο για να δούμε πώς το σύστημα μπορεί να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί. Βάσει πραγματικών περιστατικών και γεγονότων για να έχει την πλήρη του νομιμοποίηση. Um... Λοιπόν, για να συνοψίσω, ε, οι μεταβατικές αυτές αποζημιώσεις δεν θα πρέπει να είναι κίνητρα για να μην αναλαμβάνει κανείς νέα καθήκοντα. Θα πρέπει να εφαρύνουν μάλλον πρώην αξιωματούχους να βρουν δουλειά. Και επίσης η έλεγχοι και οι ε, διασταυρώσεις θα πρέπει να γίνονται πραγματικά για να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα αυτών των αποζημίωσεων. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όσους εργαστήκατε ε, στην εκπόνηση και τη δημοσίευση αυτής της μελέτης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή βάση με γεγονότα και στατιστικές για να κάνουμε τις συζητήσεις μας για την μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού, των μεταβατικών αποζημιώσεων. Σήμερα έχω την ευκαιρία και θα το κάνω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια ιδέα για το πώς το αξιολογούν το θέμα αυτό, το θεωρούν σημαντικό, έχουν σκεφτεί να το αναθεωρήσουν γενικότερα και ειδικότερα τώρα αφού ακούσαμε τις αφέστατες συστάσεις της μελέτης, το επόμενο ή τα επόμενα βήματα ποια θα είναι που μπορούμε να προβλέψουμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε οι συντάκτες, αλλιώς να δώσω το λόγο στους συναδελφούς. I think, um, what we would... Ναι, ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ε, τονίσουμε, το είπε και ο Χρήστοφ Ντέμκε, ότι χρειαζόμαστε γεγονότα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πολύ δημιουργικοί. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα εμπειρίες στα διάφορα κράτη-μέλη που μεταρρύθμισαν το σύστημα αυτό ε, προς τη θετική κατεύθυνση για τις μεταβατικές αποζημιώσεις και να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις ανάγκες αλλά να υιοθετούν και ιδέες όπως είπε ο κύριος Ντέμκε η εκπαίδευση η ε, βοήθεια, coaching ε, των πρώην μελών ή των πρώην αξιωματούχων ε, για να βρουν μια νέα δουλειά, η ομαλή μετάβαση. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ε, μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος αυτή η εμπειρία για να εμπλουτίσει και το σχεδιασμό, τη σχεδίαση μάλλον οποιοδήποτε νέου συστήματος στα θεσμικά όργανα. Η Πρόεδρος. Θέλω να δώσω την ευκαιρία μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει. Καλώς όριζω θερμά τον κύριο Πινιώτση, τον κύριο Μπουραγέ και τον κύριο Λίντρα από τη Γενική Γραμματεία. Παρακαλώ να μας πείτε και σε ποιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ε, στον κανονισμό συμμετείχε 2016 κάθετος 300 τα οποία αποφασίστηκαν πίσω από την πλάτη μας ή τη δικιά μου τουλάχιστον γιατί εγώ δεν είχα ιδέα. Κύριε Σλίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου του 2016 βασίζεται στην διάταξη της συνθήκης που δεν προβλέπει δικαίωμα πρωτοβουλία για την Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για κανονισμό που υιοθετεί το Συμβούλιο με δική του πρωτοβουλία. Χωρί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω αυτό να απαντά την ερώτησή σας. Και φυσικά έχουμε και τα άλλα νομικά μέσα που αναφέραμε που τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ε, ξέρετε, τη νομική βάση για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλα σχόλια για τη μελέτη. ε, όλοι κοιτάνε το έδρανό τους έτσι, με κάποια δυσκολία. Το ήξερα ότι θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Διαβάζοντας τη μελέτη μια-δυο φορές προσεκτικά σκέφτηκα ότι δεν θα με εκπλήξει κάτι σε αυτή τη συνάντηση αλλά τώρα πρέπει να πω έπρεπε να το είχα σκεφτεί καλύτερα. Πρέπει να πω ομιλώντας ε, εκ μέρους μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ότι αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν κατηγορώ φυσικά την ε, Κομισιόν, δεν είναι δικό σας λάθος σε καμία περίπτωση. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι αν κατάλαβα καλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κανείς δηλαδή σε αυτή την αίθουσα ούτε στον Περλεμό ούτε πουθενά σε αυτή την πόλη δεν μπορεί να κάνει κάτι για όλο αυτό με άλλα λόγια, πραγματικά ελπίζω να μην βλέπουν ε, την απευθεία μετάδοση τώρα πάνω από πέντε άνθρωποι, διότι πραγματικά αυτό είναι απίστευτο. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε σήμερα. Εντάξει, τι να πω, αλλά Πώ θα απαντήσω εγώ τις ερωτήσει δημοσιογράφων που ενδιαφέρονται για αυτή τη μελέτη και πώς θα τους πω ότι ξέρετε, συγγνώμη, αλλά προσπαθήσαμε να θέσουμε το ζήτημα και ούτως πράξαμε, αλλά μας απάντησαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ωραία, καλό είναι που υπήρξε μια μεταρρύθμιση το 2016 ε, ώστε να έχει κάπως νόημα από τους 36 ε, μήνες να πάμε στους 24, να υπάρξουν κάποια βήματα στο σύστημα, να βελτιωθούν και κάποια έλεγχη, ε, όχι μόνο η έλεγχη, αλλά τουλάχιστον να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο σαφή για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά... Αλλά όλα αυτά που αναδεικνύονται ως αδυναμίες του συστήματος ε, από τη μελέτη, πώς θα τα απαντήσουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ ότι έχω καταλάβει σωστά. Λάθος. Ότι έχω καταλάβει λάθος, συγγνώμη. Ο συνάδελφος Τάραντ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Μπλούμαγερ και κύριε Ντέμκε. Πολύ καλή αυτή η έρευνα για ένα σημαντικό θέμα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με την απόλυτη επεσιοδοξία του κυρίου Σάβαρμα απέναντι στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Συζητούμε την έκθεση αυτή, τη μελέτη και να προτείνουμε το μεγαλύτερο εμπόδιο στο δρόμο μας. Ποιο είναι. Είναι κάτι που έχω μάθει ότι λέγεται συμφωνία κυρίων. Και στη γλώσσα μου αυτό με θερμινευόμενο σημαίνει ότι το ένα θεσμικό όργανο δεν χώνει τη μύτη του στις δουλειές του άλλου. Αλλά επειδή τους έχω δει αυτούς τους κυρίους, έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, ε, κατά πόσο ντρέπονται να τις κοινοποιήσουν. Λοιπόν, αν αρχίσουμε να επικρίνουμε τις δικές μας συμφωνίες στο Κοινοβούλιο και τις αλλάξουμε, γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε, θα έχουμε και ηθικό δικαίωμα να απαιτούμε από άλλους να κάνουν το ίδιο. Είτε είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε το Ελεκτικό Συνέδριο, είτε το Συμβούλιο. Δύο παραδείγματα να σας δώσω, που είναι πραγματικά γελία. Και μήπως δεν θέλει να εξηγήσει ο κύριος Ζαβάρμα σε Πρόσφατα στην Εστονία, την πατρίδα μου, εκλέξαμε πρόεδρο, αρχηγό του κράτους, πρώην μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία κυρία εξακολουθεί να παίρνει επί μία εξαετία κάποιο είδους μεταβατική αποζημίωση για να την αποζημιώνουν που είναι αρχηγός ενός φτωχού κράτους για ποιο λόγο η πρόεδρος της Εστονίας, ανέκδοτο είναι αυτό, άνεργη είναι. Αυτό είναι υπερβολικό μέτρο και θα πρέπει οπωσδήποτε να τερματιστεί αμέσως. Όπως το κάναμε ε, το το ε, θέμα του ελεκτικού συνεδρίου που τα 28 μέλη του ελεκτικού συνεδρίου έρχονται ε, κάθε φορά, μια φορά το χρόνο για να χειροκροτούν τον πρόεδρο τους λένε. Το δεύτερο παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τους επιτρόπους υπάρχει εκεί ένας κανόνας που λέει ότι ε, για μια περίοδο που λέγεται cooling down, cooling κάτι, cooling up, εν πάση περιπτώσει για να προσαρμεστούν. Τι είναι πυρηνικό αντιδραστήρας που πρέπει να κρυώσει, αφού είσαι επίτροπος πρέπει δηλαδή λίγο να κουλάρεις. Να σας πω λοιπόν, για να πιάσεις δουλειά σε μια ιδιωτική εταιρεία, δηλώνεις το εισόδημά σου και μειώνεται η μεταβατική αποζημίωση. Και εξ όσων γνωρίζω, πολλοί επίτροποι, ιδιαίτερα από ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, ε, αποφεύγουν να το δηλώσουν. Και όταν τους το ζητήσει κάποιος ευρωβουλευτής ή τους ρωτήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαντά τουλάχιστον στην ουσία. Και τα ποσά μπορεί να είναι μικρά, αλλά παρόλα αυτά αυτό συνιστά παραβίαση των ίδιων των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ίδια έχει επιβάλει στον εαυτό της. Και οι νομικές υπηρεσίες μου είπαν να το θέσω αυτό το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όπου δυστυχώς προείδρευε πρώην Επίτροπος, η οποία αγνόησε αυτό το αίτημα και εξακολουθεί να το αγνοεί. Άλλο παράδειγμα, όπου εμείς στο Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να δράσουμε, να μην τα αγνοούμε αυτά. Το ξέρω ότι μας φέρνουν σε δύσκολη θέση, αλλά ε, ας τη ζήσουμε αυτή τη δυσκολία, να περάσουμε από αυτές τις συμπληγάδες και να προχωρήσουμε. Και τέλος, επειδή δεν συμμερίζομαι παραπάνω την απεσιοδοξία του κύριου Σαφαρμά, είναι Ηράκλειος άθλος να αλλάξουμε τις συνήθειες που έχουμε και τα συστήματα, αλλά θέλω να επενέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον για το εξή ένα, σπανίως έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, οι δικές μας μεταβατικές αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ λογικές, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, μέχρι να βρει ο πρώην Ευρωβουλευτής άλλη δουλειά και να φύγει ε, από το στρες, από τη ματέωση του να μην έχεις επανεκλεγεί ή ότι άλλη στεναχώρια και βάσανο έχεις. Στο δικό μου Εθνικό Κοινοβούλιο αυτό λύνεται με τρόπους πάρα πολύ πιο άσχημους. Όταν γίνεται ανασχηματισμός της κυβέρνησης και επανέρχεται κάποιος ε, στο βουλευτή, ως βουλευτής και φεύγει από τα ορεινά έδρανα ο αντικαταστάτης, πληρώνονται μέσα σε μισή ώρα το σύνολο του ποσού που του αναλογεί και μετά από μια-δυο μέρες, αν ξαναγίνει ένα σχηματισμός και επανέλθει στο κοινοβούλιο, δεν επιστρέφει ποτέ τα χρήματα. Εμείς είμαστε πιο πονηροί. Ε, τουλάχιστον αυτό το λάθος δεν το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Yeah, Δεν θα το σχολίαζα. Uh, uh, you might have an interest. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα και για μας ε, και θα είναι πολύ επικαιρό και στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα μετά το Μάρτιο του 2019 αναμφίβολα πολλοί κόσμος ε, και μεγάλο μέρος του τύπου θα εστιαστεί στις μεταβατικές αποζημιώσεις ε, για τους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου όταν τελικά αναχωρήσουμε. Το τελικό πρόβλημα με αυτό όπως υπόθηκε είναι ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς έρευνες ούτε υπάρχουν επαρκείς στοιχεία υπάρχει κίνδυνος ε, για γενικεύσεις. Ε, αυτό που αναφέρεται στη σελίδα 8 λέγεται ότι υπάρχουσα έρευνα υπενίστε ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε την οικονομική ανασφάλεια αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι υποζημιώσεις για διάφορους λόγους άλλους πλην της οικονομικής ανασφάλειας. Μετά τις εκλογές του 2014 κάποιοι συναδέλφοι που δεν επανεκλέγησαν δούλεψαν μόνο για πέντε χρόνια και δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά. Και αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειε του τεράστια οικονομική ανασφάλεια. Οπότε πρέπει να προσέχουμε να μην γενικεύουμε τις, τα ε, πράγματα, τι ερμηνείε, γιατί υπάρχουν κάποιοι από φτωχό υπόβαθρο και έρχονται να δουλέψουν για πέντε χρόνια με μια πενταετή σύμβαση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε αυτού του ανθρώπου. Και το τελευταίο, αν κοιτάξουμε τα νούμερα ε, στις επόμενες σελίδες. Φαίνεται ότι η σχέση με άλλα θεσμικά όργανα με μεταβατικές μας αποζημιώσεις δεν, το, δεν διαρκούν τόσο πολύ όσο άλλων και τα νούμερα δεν είναι τόσο ψηλά. Οπότε παρότι εστιαζόμαστε πολύ στους πολιτικούς θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στα άλλα θεσμικά όργανα σε, άλλα, σε άλλους εξωματούχους οπότε Ουσιαστικά αυτό πρέπει να κάνουμε τελικά είναι να έχουμε κάποια εναρμόνιση, να προσέξουμε πριν εξάγουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα. Ναι, ωραία. Αλλά θα πρέπει κάπως να έχουμε πλήρη ε, υπολογισμό. Ε, είπατε και γιατί να, να υπάρχουν καν ε, μεταβατικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι ριζικό. Αλλά μετά, όταν βρει κάποιο δουλειά, είτε είναι στο δημόσιο τομέα, είτε στον ε, ιδιωτικό, θα πρέπει να συμψηφίζεται αυτό, να αφαιρείται. Ε, στη Γερμανία είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Στην Ευρώπη δεν γίνεται. Ε, και με όλα τα υπόλοιπα είναι και θέματα συντάξεων. Υπάρχουν κάποιοι αξιωματούχοι που 30-40 χρόνια είχαν δημόσια αξιώματα και έχουν και αξιώσεις και δικαιώματα κατοχυρώσει ε, για ε, σύνταξη. Και ο κύριος Τσέλερ ε, τα, έχει αυτά τα θέματα για την απαλλαγή. Χαίρομαι που έχουν έρθει τρει εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είστε εδώ παρόντε τρει και σιωπείτε και οι τρει. αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Περιμένατε ότι δεν θα το μάθαινε κανείς. Και με το κοινοβούλιο, γιατί δεν προσπαθήσατε να βρεθεί μια λύση συνενετική και να πούμε ότι όλα αυτά τα κάναμε για τον ΑΒΓ. Φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, να μην ε, αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Και ε, Μας λέτε ότι τα αποφασίζει μόνο του το Συμβούλιο. Από πότε τα αποφασίζει μόνο το Συμβούλιο. Η διαδικασία πραγματικά βλάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της στα μάτια των πολιτών και θα έχει και συνέπειες και λυπάμαι πάρα πολύ. Και όλοι διαβάζουν στις εφημερίδες ότι εγώ θα πάρω 300.000 αποζημίωση. Δηλαδή είναι πιο ελκυστικό και πιο κερδοφόρο και συμφέρει πιο πολύ να μην επανεκλεγεί. Α, τώρα ζεστάθηκε ο κύριο Λίντρα από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Η συνθήκη είναι αυτή που είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο θεσμικό όργανο δεν έκανε πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο δεν έχει ε, εγκρίνει κανένα σχέδιο ε, ε, που ενδεχομένω να ήταν στην Τράπεζα Συζητήσεων του Συμβουλίου. Οπότε δυσκολεύομαι να δεχθώ την κατηγορία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται έχει κάνει κάτι ε, κακό ή συγκαλύψει. Εντάξει, ε, το παίρνω πίσω λέει η Πρόεδρος, αλλά από το Συμβούλιο ποιο να καλέσουμε εδώ πέρα, να κλητεύσουμε κιόλα. Ποιο είναι. Δεν μπορώ να σας πω πώς ε, ήταν η διαδικασία στο Συμβούλιο, αλλά φαντάζομαι η εκάστοτε Προεδρία παίζει ένα σημαντικό ρόλο που με βάση τις συζητήσεις που γίνονται ε, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου παίρνει πρωτοβουλία για αλλαγή. Μπορούμε να σας παρακαλέσουμε να μάθουμε ποιος είναι με τα λόγω πρόσωπα που το έχουν υποβάλει. Και ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος άνθρωπος, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο αρμόδιος. Καλό θα ήταν να μας βοηθήσετε αν δεν μας βοηθήσετε, τι να σας πω, θα, με λυπήσει πολύ. Το σημειώνω και θα επανέλθουμε με απάντηση. Ε, μήπως να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει άλλη πρωτοβολία που είναι η μεταρρύθμιση του κώδικα συμπεριφοράς και δεντολογίας των επιτρόπων που παρουσίασε ο πρόεδρος Ιούνκερ το Σεπτέμβριο στη ε, συνεδρίαση της Ολομέλειας για την κατάσταση στην Ένωση και τώρα τον έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένει την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Και ένα από τα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης είναι η ε, παράταση της περίοδου cooling off από 1,5 χρόνο σε 2 και δεν ισχύει η διαφάνεια, ενώ για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3 χρόνια εκεί που μπόρεσε κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλαβε την πρωτοβουλία και συμβουλεύτηκε το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο. Όντως, έχουμε κάνει και πολλές άλλες προτάσεις για το τι άλλο θα μπορούσατε να είχατε κάνει. Θέλω να δώσω το λόγο κατ' εξαίρεση σε εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών από τη διεθνή διαφάνεια λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Από την απόψη μας, διαφάνεια, διεθνής διαφάνεια, το πιο σημαντικό είναι βέβαια να αποφεύγονται τα, οι συγκρούσεις συμφερόντων όταν εξωματούχοι περνούν από τη, μία τους, από τη θητεία τους σε κάποια άλλη απασχόληση. Ε, μάλιστα έχουμε κάνει μια μελέτη που δημοσιεύσαμε φέτος τον Ιενάρη, όπου αναλύουμε τη διαδρομή όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στη διάρκεια της τελευταίας θητείας που έχουν φύγει πια από την Ένωση. Ε, και είδαμε ότι η σταδιοδρομία 500 ανθρώπων, ε, το 1 τρίτο εξ αυτών παραμένουν σε κάποια δημόσια ε, υπηρεσία από την εθνική τους αρχική εντολή ή άλλες θέσεις κατέχουν, το 1 τρίτο φεύγουν από το εργατικό δυναμικό ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για το τι είδους απασχόληση έχουν και το 1 τρίτο εξ αυτών πιάνουν νέα δουλειά. Ανάμεσα στο 1 τρίτο αυτών βρίσκουμε ότι το 100 των πρώην Ευρωβουλευτών ε, απασχολούνται από ε, λόμπι τα οποία είναι γεγραμμένα στον κατάλογο των λόμπι της Ένωσης. Συστημικό ζήτημα λοιπόν εδώ, όπου μπορεί όντως να υπάρχουν και να προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων όταν ε, οι ξεματούχοι φεύγουν από την θητεία τους, τελειώνουν τη θητεία τους. Δεν έχουμε ένα περιορισμό μετά από την απασχόληση για τους ευρωβουλευτές, πράγμα που είναι πολύ παράξενο δεδομένου ότι ε, το προσωπικό που υποστηρίζει αυτούς τους ευρω... ίδιους ευρωβουλευτές ε, έχουν ε, περιορισμούς όταν σταματάει να είναι μέλος του υπαλληλικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το καταστατικό που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Πρώτου, ζητείται κοινοποίηση από πλευρά των Ευρωβουλευτών να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τη θέση που θα κάλυψουν όταν θα φύγουν. Βλέπουμε ότι το στοιχείο κλειδί εδώ είναι, εφόσον όλες αυτές οι υποθέσεις είναι, σε όλες αυτές οι υποθέσεις είναι να εντοπίσουμε αν υπάρχει όντω σύγκρουση συμφερόντων όταν ένας άνθρωπος φεύγει από εδώ, ένας βουλευτής φεύγει από εδώ και απασχολείται από έναν τομέα όπου προηγουμένως ε, νομοθετούσε. Χρειάζεται ανεξάρτητος έλεγχος και εποπτεία. Αυτό είναι αλήθεια για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι θεσμοί είναι οι ίδιοι που θεσπίζουν τους κανόνες για τη μεταβατική αποζημίωση και την απασχόληση των ε, μελών τους μετά και μετά ε, βλέπουν οι ίδιοι αν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο γίνεται και με τους επιτρόπους. Αυτοί είναι που επιβλέπουν αν οι πρώην του συνάδελφοι ή οι προκάτοχοι ε, κάνουν κάποια ε, και τι, ποια και τι δουλειά κάνουν, ενώ για τους ευρωβουλευτές δεν υπάρχει καν εποπτεία. Κάποιες διεθνείς μελέτες λοιπόν δίνουν κάποιες ιδέες για το τι είδους ε, στοιχεία θα έπρεπε εδώ να λαμβάνονται υπόψη. Να πω ότι ε, η επίσημη οι επίσημοι κάτοχοι αυτών των αξιωμάτων πρέπει να ενημερώνουν στο Καναδά και στην Γερμανία ας πούμε από τον, ε, την Καγκελάριο ε, δίνεται ένα σχέδιο μετά ας πούμε, ε, δεν μπορεί να, να, να, να, εγκρίνει το σχέδιο για έναν αγωγό και μετά να προεδρεύει στην εταιρεία που κατασκευάζει τον, προεδρε... τον αγωγό αφού έχει λήξει η θητεία του. Ε, είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει πολλά για αυτή την κατάσταση, μπορεί να κάνει ε, πολλά και να ε, τονίσει ποια είναι η κατάσταση, καθώς και να ζητήσει αλλαγές πολλές από αυτές τις πτυχές ε, που ορίζονται Ορίζονται και προβλέπονται και μηχανισμοί οι οποίοι βελτιώνουν την κατάσταση. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στο σύστημα είναι ότι το μάκρος της μεταβατικής αποζημίωσης συνδέεται με το μάκρος της υπηρεσίας. Ε, και αυτό έχει νόημα. Θα πρέπει να το κάνουν και άλλοι θεσμοί. Ε, τώρα αυτό που δεν κάνει όμως το Κοινοβούλιο και που το έχουν άλλοι θεσμοί είναι ότι αν ξεκινήσεις μια νέα δουλειά σε τον ιδιωτικό τομέα αυτό το ποσό αφαιρείται από τη μεταβατική, ε, τη μεταβατική αποζημίωση, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί κατεπηγόντως, όπως είπε και κάποιος από το Προεδρείο. Μάλιστα. Αναμένουμε. Τριακόσια... 216. Δεν ξέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ρυθμιστεί αυτό και μετά τις τελευταίες ε, ευρωεκλογές ε, κάπως ευθυγραμμίστηκαν αυτά με τους μισούς των ευρωβουλευτών, των επιτρόπων. Αλλά έπρεπε να το συγκρίνουμε με το τι γίνεται στα κράτη-μέλη και πώς συμψηφίζονται αυτά τα ποσά. Κρίμα. Έχουμε πολλή δουλειά. Ο συνάδελφος Σάβαρμα, θέλετε να τοποθετηθείτε και πάλι οι συντάκτες Εν συντομία, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ αργά ή γρήγορα κάποια στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου θα αποτελέσουν αντικείμενα κριτικής προς τους αξιωματούχους. Ο λόγος που αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις μεταβατικές αποζημιώσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά αργά ή γρήγορα θα ενταθεί το ενδιαφέρον και θα, θα γίνουν προσπάθειες ανάλυσης του κανονιστικού πλαισίου, θα τεθούν ε, ερωτήματα νομιμοποίησης των ε, πληρωμών αυτών και θα αρχίσουν επικρίσεις. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Όσον αφορά την οικονομική ανασφάλεια, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ναι, φυσικά υπάρχουν πολιτικοί και αξιωματούχοι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μετά από το πέρας της υπηρεσίας τους. Ελάχιστες ερεύνες έχουν γίνει επί του ζητήματος αυτού, διότι ε, παρεμβαίνει και σε ζητήματα ιδιωτικού απορρίτου. Αλλά η όποια έρευνα έχει γίνει μέχρι στιγμής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα οικονομικά προβλήματα ε, αφορούν μόνο ελάχιστους αξιωματούχους Στη μελέτη μας λοιπόν έχουμε κάνει και προτάσεις και για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, φυσικά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι αξιωματούχοι πολιτικοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν ε, οικονομικέ δυσκολίε μετά το πέρα τη θητεία του, οπότε γιατί να μην του καταβληθούν μεταβατικέ αποζημιώσεις εφόσον υπάρχει ανάγκη. Εμεί συμφωνούμε με αυτή την σύσταση, αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βασιστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτό τον ισχυρισμό, ότι πρέπει να βοηθήσουμε κάποιου ανθρώπους ε, για τι οικονομικέ δυσκολίε που ενδεχομένω θα αντιμετωπίσουν αφού είναι τόσε λίγε, περιπτώσει. Αυτό είναι που μα δημιουργεί πρόβλημα. Ευχαριστώ, συνάδελφο, ο Σαβάρμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να συνοψίσουμε να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να διορθώσω τον κύριο Ταράγγεν. Σπάνια πρέπει να τον διορθώσω, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνω. Δεν είναι μόνο θέμα απεσιοδοξίας. Ε, αναφέρομαι και στην Transparency International. Ευχαριστούμε κύριε Τάραντ μάλιστα που μου ξαναδώσετε πίστη στο ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο. Να διορθώσουμε την απόφαση του 2005. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι και πυρηνική φυσική. Είμαι βέβαιος ότι το 90% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποια σφάλματα τα οποία υπάρχουν ακόμα. Την ημέρα υπαριθμών 1, αφού κανείς αποχωρήσει από εδώ, όταν φύγω εγώ από εδώ, αν βρω μια νέα δουλειά, αν καταφέρω να βρω μια νέα δουλειά, γνωρίζοντα ότι είναι πολύ πιθανό να μην επανεκλεγώ ή για οποιονδήποτε λόγο. Και εφόσον λαμβάνω μισθό από αυτή τη δουλειά, την ημέρα μετά από την ημέρα, τη μεθεπόμενη, εφού αποχωρήσω από εδώ, γιατί να ε, πάρω 7, 8, 12 μήνες αποζημίωση. Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά αυτό είναι μόνο μια πτυχή του ζήτηματο. Αυτό που με απελπίζει περισσότερο είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει επαρκής διαφάνεια σε περιπτώσεις όπου για παράδειγμα είχαμε έναν επίτροπο που υπήρξε επίτροπος για ελάχιστου μήνες ή κάποιος που υπηρέτησε για ένα χρόνο στα θεσμικά όργανα για δύο και μετά ξαφνικά παίρνει ε, ένα σώρο λεφτά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ορισμένε περιπτώσεις. Αυτό, ούτε αυτό είναι πυρηνική φυσική. Κάποιος πρέπει να το φτιάξει όμως αυτό. Κύριε Βόν, συμφωνώ μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι τόσο εύκολο για τους πολιτικούς να βρουν μια νέα δουλειά σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε σε γενικές γραμμές καλό είναι να μην λέμε ότι ισχύει το ίδιο για όλους. Και εγώ γνωρίζω μια περίπτωση σε ένα θεσμικό όργανο όπου ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος βρέθηκε άνεργος για σχεδόν τώρα δύο χρόνια από τότε που αποχώρησε. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες περιπτώσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να δούμε το κανονιστικό πλαίσιο και να το επιδιορθώσουμε. να έχουμε ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο βασισμένο σε γεγονότα, σε αυτά στοιχεία. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, μια πρόταση, κυρία Γιάλα Σέντερ, συμφωνώ πολύ. Γιατί έχω υπόψη μου διάφορες περιπτώσεις που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, ούτε επίδομα ανεργίας δεν παίρνει. Μετά από δύο και τρεις θητείες ε, ευρωβουλευτή. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες. That uh, ε, πάντως, χρειαζόμαστε τους καλύτερους. Όπως το είδαμε και για ε, τους δημοσίους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Θέλουμε τους καλύτερους. Δεν βρίσκαμε κόσμο από διάφορα κράτη-μέλη, γιατί οι μισθοί δεν ήταν τόσο ελκυστικοί όπως εκείνη στη χώρα τους, λαμβάνοντας υπόψη τον εκπατρισμό, την αποδημία και άλλα προβλήματα οικογενειακά κτλ. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις δύο πλευρές. Αν θέλουμε τους καλύτερους λοιπόν να εξασφαλίσουμε να είναι το πακέτο ελκυστικό για να έρχονται οι καλύτεροι και να ενδιαφέρονται, να προσελκύονται από αυτές τις προσφορές και αυτές τις θέσεις και τα αξιώματα Πάντως συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει όλος ο κύκλος να είναι απολύτως διαφανής. Τώρα έχουμε τη δέσμη μέτρων για τις μεταφορές όπου ο κάθε οδηγός φορτηγού υφίσταται επιθεωρήσεις εργασίας, επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολύ λιγότερους ανθρώπους που φεύγουν από σημαντικές θέσεις οι ευαίσθητες θέσεις και δεν μπορούν να ελεγχθούν με τρόπο σωστό. Που να πληρώνονται σωστά και δίκαια, αλλά όχι περισσότερο ούτε λιγότερο από ό,τι αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Πρόεδρος. Θα πρέπει να κάνουμε μία λίστα για το τι πρέπει να γίνει και να το στείλουμε αρμοδίως. Γιατί κρεμούν κάποια ζητηματάκια επιγόντως που πρέπει να ρυθμιστούν. Και μπορώ να σας αναφέρω και περιπτώσεις. Να ξέρουμε ε, πώς ε, τα ρυθμίζει αυτά η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη, πολύ ενδιαφέρουσα και για την παρουσίαση αυτής. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της πρωινής συνεδρίασης, σύντομη παρουσίαση πρόσφατα δημοσιευμένης ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδική έκθεση 15 του 17, εκ των προτέρων αρισιμότητα και αποθεματικό επίδοση στη συνόχη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Καλωσορίζω τον κύριο Μπάλκο που θα μας την παρουσιάσει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι για να προσανατολιστούμε περισσότερο προς τα αποτελέσματα ε, έχουμε φτιάξει την εκ των προτέρων αρεσιμότητα και το αποθεματικό επίδοσης. Ε, σε άλλους ελέγχους έχουμε εξετάσει κατά πόσο αυτές οι πολιτικές όντως έχουν δώσει καλύτερα κίνητρα ε, ή όχι. Υπάρχει πραγματική καινοτομία και κατά τη γνώμη μας παρέχεται ένα συνεπές πλαίσιο ώστε να εκτιμούμε την ετοιμότητα των κρατομελών ώστε να εφαρμόσουν τα ε, κονδύλια στη, κατά την προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, η Κομισιόν εκτιμώντας τις ερεσιμότητες δεν έλαβε υπόψη ε, ε, τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, πληροφορίες που παίρνουμε από τη Γενική Διεύθυνση, από τις δικές μας ε, δραστηριότητες παρακολούθησης. Έχουμε παραδείγματα ασυνέπειας που δείχνουν και έλλειψη θένους όταν, όταν πιστοποιούμε την αυτό, ε, αξιολόγηση. Ήταν εξαιρετικά θετική και εξαιρετικά και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αποτηρώνται οι αιρεσιμότητες γιατί εν γέννη υπάρχει χώρος για ερμηνεία. Ε, επίσης δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι αιρεσιμότητες επηρεάζουν τις αλλαγές επιτόπου ή θα οδηγήσουν σε αλλαγές επιτόπου, πράγμα που είναι και ο τίτλος της ειδικής μας έκθεσης σε πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων δράσης, τα κρατημέλη έχουν δεχτεί να τηρήσουν ε, τους επιπλέον όρους, ενώ η Κομισιόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να αναστείλει πληρωμές σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων. Επιπλέον, μετά από την υιοθέτηση των προγραμμάτων, η Κομισιόν δεν προβλέπει την αναστολή πληρωμών πριν από την εξεκθέση των των μελών για την ολοκλήρωση των δράσεων για την ε, τήρηση των όρων. Ε, κατά τη γνώμη μας, ε, ε, θα πρέπει να συμβάλλουν όλα αυτά στην καλύτερη χρήση των προγραμμάτων των project, ώστε να μην έχουμε ε, λίγο στα αποτελέσματα. Πολύ συχνά οι πληρωμές καταβάλλονται ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρωση οι στόχοι μέχρι την τέλος προθεσμίας του 2018. Οι αναστολέ και οι οικονομικές διορθώσεις για την υποαπόδοση είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπόκειται σε πολύ περιοριστικές όρους Επί τη βάση των ελέγχων μας δεν πιστεύουμε ότι οι ρυθμιστικές αλλαγές των δύο μέσων στη διάρκεια της περίοδου θα είναι αποτελεσματικές ε, σε σχέση με το κόστος τους. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στις συστάσεις, ε, μία σειρά συστάσεων για καθένα εκ των δύο μέσων εφόσον αυτά διατηρηθούν. Εάν ναι θα πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε να είναι πιο να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική χρήση των δαπανών για τη συνοχή. Το πρώτο σύνολο συστάσεων ε, εστιάζουν στις εξάντε ε, ερεσιμότητες για την περίοδο μετά το 2020. Λοιπόν, η Κομισιόν θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις ερεσιμότητες ως μέσο για να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις ε, ε, καταβολές και να τηρήσουν τις αιρεσιμότητες ε, ε, διατηρώντας όμως μόνο τις αιρεσιμότητες που οδηγούν στην πραγματική εφαρμογή και επίτευξη των στόχων των πολιτικών. Δεύτερον, να συμβαδίζουν με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, τρίτον, κοινή συνεννόηση του τι πρέπει να επιτευχθεί και τέλος να πετήσουν την πλήρωση και την εφαρμογή των όρων στη διάρκεια ολόκληρης προγραμματικής περίοδου. Το δεύτερο και τελευταίο σύνολο συστάσεων εστιάζεται στο αποθεματικό επίδοσης. Εμείς πιστεύουμε πως η Κομισιόν θα πρέπει αυτό να το μεταβάλει σε ένα ε, μέσο το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και θα χορηγεί δηλαδή κονδύλια σε όσους πετυχαίνουν τα καλά αποτελέσματα. Τα δύο τρίτα δηλαδή να βασίζουν... να αφορούν ε, την καλή απόδοση, όπου όμως ε, οι project managers θα πρέπει να αποδείξουν τι θέλουν να επιτύχουν με αυτή την επιπλέον χρηματοδότηση, έπειτα να μετα, δούμε τα βήματα εφαρμογής με στόχο την καλύτερη απόδοση μακροπρόθεσμα για τις συγκεκριμένες υποδομές και τέλος να αναθεωρηθούν οι όροι προς την αναστολή και τη διόρθωση ώστε να μπορούν, μπορεί η υποαπόδοση να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου κύριε και κύριοι, η Κομισιόν καλωσορίζει την ειδική εκθέση για τις εκ των προτεραιών και το πλαίσιο επιδόσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου στην περίοδο 2014-2020 οι αιρεσιμότητες και το αποθηματικό επιδόσεων έδωσαν κίνητρα για καλύτερες δαπάνες, απαιτώντας από τα κράτη-μέλη να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσει του σχεδιασμού και την υλοποίηση των κονδυλίων. Η έκθεση συνιστά όλα τα μέσα εφόσον διατηρηθούν να ενισχυθούν μετά το 2020. Η Κομισιόν γενικά εγκρίνει τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου τονίζοντας ότι για τις μελλοντικές προτάσεις δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ε, εκφράσουμε κάποια θέση. Όσον αφορά τις εκ των προτεραιών αιρεσιμότητες ή προϋποθέσεις για επιτυχείς επενδύσεις, είναι κάτι καινούριο στην πολιτική συνοχής αφορούν συγκεκριμένου ε, τομεί ε, με συγκεκριμένε προϋποθέσεις για κονδυλία και χρηματοδότηση από τα διευθυντικά και επενδυτικά ταμεία. Αυτές οι εκ των προτεραιών αρεσιμότητες ε, έχουν ε, αποκτήσει τεράστια επιρροή συνεισφέροντας στη βελτίωση του γενικού επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάρτιο φέτος η Κομισιόν δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασία για την προστέμινη αξία των εκ των προτεραιών αρεσιμοτήτων στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Έδειξε η μελέτη αυτή ότι παρήχαν ε, κίνητρα στα κράτη και στις περιφέρειες για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πολιτικές και ειδικότερα στο πλαίσιο των συστάσεων κατά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 36 είναι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αφορούν τα ταμεία του, ε, της πολιτικής συνοχής. Ορισμένες είναι γενικής ε, φύσης, όπως ε, δημόσιες συμβάσεις, ε, κρατικές ενισχύσεις και 29 είναι θεματικές. Σχετίζονται με συγκεκριμένες ερεσιμότητες ε, τομέων σε τομείς που υποστηρίζονται την πολιτική συνοχή. Περίπου το 75% τα τρία τέταρτα αυτών των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είχαν εκπληρωθεί τη στιγμή υιοθέτηση των προγραμμάτων. Όπως αναφέρθηκε ήδη από το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, Ε, δημιουργήθηκαν πάνω από 700 σχέδια δράσης. Μη ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων δράσης είναι λόγος αναστολής πληρωμών από την Κομισιόν. Μέχρι σήμερα μόνο το 2% αυτών των σχεδίων δράσης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες η Κομισιόν θα εκπονήσει την τελική της γνωμοδότηση για τα υπολοιπόμενα σχέδια δράσης και θα αποφασίσει αν θα αναστείλει τις πληρωμές ή όχι. Τώρα, για το αποθεματικό επίδοσης ε, και το σχετικό πλαίσιο, όπως ξέρετε, έχει συμπεριληφθεί στα προγράμματα ε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις μικρομεσαίες και της τεχνικής αρρωγής αφορά συγκεκριμένους δείκτες ε, επιδόσεων και αποτελεσμάτων που πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2018 και στόχου ηχή που πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2023. Τα επιτέγματα θα αξιολογηθούν το 2019 από την Κομισιόν. Αυτή η αξιολόγηση θα αποτελεί τη βάση για την ε, εκχώρηση του αποθεματικού επίδοσης που είναι 6% πρόσθετο κονδύλιο που μπορεί όμως ε, να οδηγήσει και σε αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών σε περίπτωση σοβαρών υποεπιδόσων. Η επίτευξη των στόχων θα αξιολογηθεί ξανά το 2020 και σε περίπτωση πολύ χαμηλών επιδόσεων μπορεί να ε, υπησέλθουν οικονομικές διορθώσεις. Η αναθεώρηση ε, των επιδόσεων το 2019 θα γίνει κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ε, επίδοση και τα αποτελέσματα και την υλοποίηση των βασικών βήματων. Τέτοιοι δείκτες επηρεάζονται απευθείας από τους διευθυντές του προγράμματος και συνδέοντας τα επιτέγματα με τρόπο σαφή και μετρήσιμο. Ο μηχανισμός αυτός αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο σχεδιασμού πρόβλεψης των προβλημάτων και αντιμετώπισης τους. Βοηθά επίσης τις διαχειριστικές αρχές να εστιαστούν στους κύριους στόχους πολιτικής. Συμβάλλει μαζί με άλλα ε, στοιχεία το ίσως προσανατολισμό για τις επενδυτικές ανάγκες, ε, τη λογική των σαφών στόχων και δικτών στα κριτήρια επιλεξιμότητας, ε, στην επίτευξη των στόχων μέσω μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής υποστήριξης θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και τέλος εστίαση της επιδόσεις και μεγαλύτερη σύνδεση με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά μας απασχολούν στο επίκεντρο της μελλοντική πολιτικής. Τα πολύτιμα σχόλιά σας και η υποστήριξή σας θα μας βοηθήσουν και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ε, για αυτό τον έλεγχο επιδόσεων. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή έκθεση πραγματικά και πολύ επικριτική έτσι. Και δείχνει ότι πώς να το πω, αποφασίζουμε τρελά πράγματα σούπερ, τα οποία όμως μετά δεν εφαρμόζονται. Και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν εφαρμόζονται πάρα πολύ κρίσιμα πράγματα της νομοθεσίας. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ο συνάδελφος Πυρίνσκι είναι ο εισηγητής, έχει μέσα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχουμε. Δεν είμαι βεβαίως ότι έχουμε πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομος. Ένα λεπτό ολόκληρο. 45 λεπτά μου φάγατε 15, ε, δευτερόλεπτα μου φάγατε τα 15. Λοιπόν, ένα θέμα που κυριαρχεί παντού, Πρόεδρε, ε, και το αναφέρατε κι εσείς, είναι αυτό που θέλω να αναφέρω. Ακούσαμε χθε την Επίτροπο Τέισεν και η συζήτηση ήταν για την υλοποίηση και την απορρόφηση των ταμείων και των πόρων. Και ένα από τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι εκ των προτέρων ερησιμότητα είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα τώρα για το ο χαρακτήρα ή τη γενική μεταρρύθμιση και δεν συμμαζεύεται. Απλώς θα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε τώρα στα σημαντικά κριτήρια ή εκ των προτέρων ερεσιμότητες και το αποθεματικό επίδοσης βοηθούν, διευκολύνουν, επιταχύνουν την ε, απορρόφηση. Η απάντηση η σύντομη είναι όχι. Εγώ δεν θέλω να απορρίψω τη συνέχιση αυτών των διευθετήσεων στην επόμενη ε, προγραμματική περίοδο. Αλλά όπως είπατε και εσείς η ίδια, και συμφωνώ για την έκθεση ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντική η έκθεση και μας οδηγεί και σε μεγάλη σκέψη. Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν και κατά πόσο και με ποια μορφή θα συνεχιστεί αυτό. Και αν είναι αυτές οι προσεγγίσεις σκόπιμο να διατηρηθούν. Ε, αναφέρομαι εδώ σε δύο παραγράφους της έκθεσης, την παράγραφο 39 και την παράγραφο 72, όπου γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι η εκ των προτέρων ερεσιμότητες. έτσι όπως έχουν αυτές καθ' αυτές, δεν σημαίνει ότι βελτιώνουν την εφαρμογή και στο 72 το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι για την προγραμματική περίοδο το 14 με 20 δεν σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα σε σχέση με παρελθούσες περιόδους. Τίθενται λοιπόν διάφορα ερωτήματα που θα ήθελα και εγώ να προσέξουμε. Τώρα δεν νομίζω να έχουμε χρόνο να εμβαθύνουμε, αλλά θα περιμένω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ελεκτικό Συνέδριο να επανέλθουν, ενδεχομένως και γραπτό σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ναι. Είναι συστημική η σημασία της έκθεσης, οπωσδήποτε θα την εγγράψουμε ξανά στην ημερήσια διάταξη. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ακριβώς ε, η μία εφαρμογή της ερεσιμότητας συνηγορεί ε, κατά της ερεσιμότητας ή κατά της εφαρμογής. Νομίζω κατά της εφαρμογής, γιατί η κατα της εφαρμογης νομιζω κατα της εφαρμογης γιατι η αρισιμοτητα και τα, ε, οι όροι και οι κανόνες είναι ορόσημο. Κύριε Μπάλκο, εκτιμάτε δυνατό, ε, ε, εκτιμάται ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί η αιρεσιμότητα μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Uh, course, uh, this is very important question, Madam Chair. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό κυρία Πρόεδρε. Κατά τη δική μου απόψη φαίνεται πολύ σημαντικό. Όπως υπογραμμίσετε και εσείς στην αρχή της παρεμβασής σας, η έκθεση αυτή είναι κρίσιμη σημασία και όπω υπογράμμισε και ο κ. Περίνης ο συζητητής ε, της Επιτροπής αυτής ε, ήταν πολύ προκλητικό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της έκθεσης αυτής ε, αξιοποιώντας και τα σχολιά σας. Ήθελα απλά να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε επικριτικοί ε, όχι μόνο σε αυτή την έκθεση. Για παράδειγμα, προετοιμάζουμε μια έκθεση εστίασης στη βιωσιμότητα για το τι είναι απαραίτητο. Εκπονούμε μια έκθεση για την απλούστευση. Ε, κάτι που, για, την, για το οποίο θα είμαι εγώ αρμόδιο. Μου φαίνεται, όπως είπατε και στην αρχή, ε, ότι ναι, η απάντηση είναι ναι, βεβαιότατα. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα επανέλθουμε Όμω, Θέλω να θυμίσω ότι στις 2.30 ε, θα, θα ξαναπούμε έχουμε μια ώρα συνεδρίαση για την έκθεση για την Ελλάδα και μετά έχουμε το τριμερή διάλογο. Λήξη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.